Okay, guten Morgen. Ich brauche ein Fernglas, um Sie... Καλημέρα. Μα θέλω κι άλλα για να σας δω. Λοιπόν, Ξεκινάει η συνεδρίαση, η έγκριση της ημερήσιας διάταξης, έκθεση Αλφονσί για τις γλώσσες που κινδυνεύουν. Αποφασίσαμε να αναβληθεί, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές ε, τροπολογίες. Ε, συμφωνείτε? Ναι. Ωραία. Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση λοιπόν το 11. Σημείο 3, 2 της ημερησίας διάταξης. Πρακτικά της 22ης 23ης Απριλίου 2013. Αν έχετε κάποια παρατήρηση παρακαλώ να το πείτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για να αλλάξουμε κάτι. Δεν έχουμε εστονικά, λιθουανικά, λετονικά, μαλτέζικα και σουηδικά σήμερα. Μετά, έχω να σα πω το Είχαμε τον το τριμερή διάλογο για τους νομοθετικούς φακέλους. Το ένα αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και αθλητισμού. Είχαμε άλλες δύο συναντήσεις από την τελευταία συνεδρίαση, 23 Απριλίου και 14 Μαΐου. Πλησιάσαμε αρκετά θα έλεγα στις θέσεις μας. Έχουμε σχεδόν συμφωνήσει στο κεφάλαιο εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός. Μπορώ να σας πω πως το Συμβούλιο μας είπε πως μπορούμε να διατηρήσουμε τα ονόματα όλων των προγραμμάτων. Έχουμε ξεχωριστό προϋπολογισμό για τη νεολαία. Αυτό σημαίνει πως επιτύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε. Και για χάρη του Συμβουλίου και επειδή κάναμε κάπως πιο στους τους στόχους μας, όλα αυτά γίνανε για να ε, συμβαστούμε και με αυτά τα οποία έκανε δεκτά το Συμβούλιο Εράσμους, Κομμένιος, Γκρούντιχ και Σπότ. Έχουμε δύο ακόμα προβλήματα. Το ένα είναι το πρόβλημα του ονόματος, του, του τίτλου του προγράμματος. Το δεύτερο είναι πως το Συμβούλιο θέλει να δει πάρα πολύ περιοριστικά το ζήτημα των ε, δανείων ε, μάστερ. Θέλει να αφιερώσει για αυτό το ζήτημα μόνο 2% του προϋπολογισμού. Η Κομισιόν ε, είχε προβλέψει ένα 5% για αυτό το κομμάτι του μάστερ και του σχετικού δανείου. Το πρόβλημα είναι πως η Κομισιόν μας λέει πως η υπόθεση αυτή μπορεί να ε, υπάρξει μόνο με μια γεωγραφική κατανομή εάν ε, έχουμε ένα τουλάχιστον 4%. Με 2% δεν γίνεται. Συμφωνούμε και εγώ προσωπικά θέλω να υπάρξει αυτή, αυτό το μέσο για δάνεια και Περίεργος αυτή τη φορά είμαστε με το μέρος της Κομισιόν ε, ενάντια στο Συμβούλιο για να αυξηθεί τουλάχιστον στο 3,8% το ποσό. Το δε Συμβούλιο με την αιτιολόγηση πως πρέπει να κάνουμε οικονομίες ε, έκοψε τον προϋπολογισμό της εκτελεστικής υπηρεσίας Κομισιόν κατά 0,2% και τα έβαλε στις εθνικές ε, υπηρεσίες. Ε, δηλαδή έτσι πάνε αυτά, άλλοι κάνουν οικονομίες και άλλοι παίρνουν περισσότερα. Ελπίζουμε να πάμε στο 3,4% και να πάει 3,4% ε, και 1,8% στην Κομισιόν. Τελικά καταφέραμε αυτά τα οποία θέλαμε. Υπάρχει ακόμα μόνο το ζήτημα του τίτλου και του μέσου δανείων. Ε, από ό,τι φαίνεται επί Ιρλανδικής Προεδρίας δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα ακόμα. Θα έχουμε ε, την αλλαγή του ονόματος και το ζήτημα το, του μέσου δανείων, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο προπολογισμό. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να το διαπραγματευτεί η Επιτροπή του Προπολογισμού και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα των πράξεων ε, κατεξιοδότηση. Αλλά αυτό είναι οριζόντιο ζήτημα. Δεν μπορώ να το λύσω εγώ. Και να ήθελα. Υποθέτω πως θα μπορέσουμε να ψήσουμε το Σεπτέμβριο τώρα πια. Μέχρι τότε θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Creative Europe. Είχαμε τον δεύτερο άτυπο τριμερή διάλογο 25 Μαρτίου. Δεχτήκαμε ένα συμβαστικό κείμενο, δεν έχουμε κανένα σοβαρό πρόβλημα. Επόμενος τριμερής διάλογος 30 Μαΐου. Για τα εκκρεμή προβλήματα ισχύει αυτό το οποίο ισχύει ε, και με τον προπολογισμό. Σήμερα βεβαίω θα ψηφίσουμε την πολιτιστική πρωτεύουσα. Και αυτό είναι θέμα συναπόφασης που πρέπει να διαπραγματευτούμε, αλλά νομίζω πως θα τελειώσει αυτό πάρα πολύ γρήγορα το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει καμία πράξη εφαρμοστική κτλ. Το πρόβλημα της ε, νηπικότητας ε, και εδώ πέρα το ζήτημα είναι τα λεφτά. Η Κομισιόν και πάλι έχει κόψει ένα 5%. Μιλάμε δηλαδή για μια περικοπή 23% σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Στο πρόγραμμα αυτό, έτσι, του, του Ευρωπαίου Πολίτη. Είναι μικρά, μικρά τα ποσά και να τα περικόψουμε μετά και κατά 23%. Εγώ απίθυνα μια επιστολή εξ ονόματός σας στον Μπέγκε, στον Λαμασούρ και λοιπούς και τους είπα να προσέχουν, δηλαδή γινόμαστε γελοί. Αλλιώ δεν μας παίρνουν καθόλου σοβαρά πλέον. Αυτά τα θετικά και τα αρνητικά και μπορώ να σας ανακοινώσω πως δεν υπάρχει καφές. Γιατί, γιατί κάνουν απεργία. Οπότε να σας εξηγήσω το εξής. Όταν συνεδριάζουμε εδώ σε αυτή την αίθουσα, έχουμε δικαίωμα σε καφέ. Πόσες θέσεις υπάρχουν εδώ πέρα? 450. Υπολογίζουν λοιπόν 450 καφέδες και τους πληρώνουν ε, όλας παρά το ότι προφανώς δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα. Θα πω το εξής λοιπόν. 850 ευρώ έτσι. Ανασυνεδρίαση. Ωραία. Ξέρω που μπορούμε να κόψουμε λεφτά λοιπόν. Εκεί πέρα. Γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι καφές αυτό σερβίρουν. Είχε έρθει ο Κόλ εδώ πέρα κάποτε και μου είπε άμα μου ξανασυμβείτε τέτοιο καφέ θα ξαναπατήσω. Στη δε Γερμανική Βουλή δεν σερβίρουν καφέ καθόλου. Ε, έχει λίγο νερό στη γωνία, εντάξει, είναι και υγιεινό. Αλλά ο, ο καφές δεν χρειάζεται. Πρώτον, δεν είναι υγιεινός. Δεύτερον, δεν έχει γεύση. Και τρίτον, είναι και πανάκριβος. Λοιπόν, μια που δεν Είχαμε καφέ σήμερα και ζούμε όλοι. Προτείνω να κάνουμε την εξή εξοικονόμηση. Να σταματήσει όλη αυτή η υπόθεση των καφέδων. Δεν ξέρω, μπορεί να με βρίσκεται κακιά, αλλά θεωρώ πως μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Δηλαδή αν κάθε συνεδρίαση κοστίζει 850 ευρώ για το τίποτα, δεν πειράζει. Α, λίγο λίγο εκεί και τελείωσε. Ευχαριστώ κύριε Μιγκάλσκι, ευχαριστώ. Οι άλλοι με στραβοκοιτάνε βεβαίως. Αλλά πραγματικά ο καφές αυτός δεν, δεν, δεν πίνεται κιόλας. Και άμα σας αρέσει, τι να πω. Λοιπόν, σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Όθηση στο του πολιτισμού και της δημιουργία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Μαρή Τερέζ Σάντσες Σμιτ. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να προτείνω αντί να έχουμε τέτοια μπουκάλια να μας βάζουν χήμα νερό. Νομίζω ότι σε αρκετά κοινοβούλια του κόσμου το νερό δεν είναι εμφιαλωμένο. Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που θα μιλήσω για τη δημιουργία σήμερα. Είχα πρωινό με τους εκπροσώπους αυτών των βιομηχανιών στην Ευρώπη και υπάρχουν κάποια πολύ θετικά σημεία και θέλουμε να προωθήσουμε τον τομέα αυτό για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση που μας απασχολούν σήμερα στην Ευρώπη. Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της για την προώθηση του πολιτιστικού τομέα Σαν μέλος αυτής της Επιτροπής λοιπόν για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση είναι τιμή μου που ε, η πολιτιστική παραγωγή είναι στο κέντρο των ε, δραστηριοτήτων μας σήμερα. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την περίοδο κρίσης. Το πολιτιστικό κομμάτι πάντα χαρακτήριζε την πολιτική μας και αυτό το αποδεικνύει αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική εξαίρεση. Η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο την προηγούμενη Πέμπτη με αφορμή την αντολή διαπραγμάτευση για την ελεύθερη ζώνη με τη ΣΥΠΑ δείχνουν το ενδιαφέρον μας για την προστασία της. Δύο τρίτα υπεψήφισαν την εξαίρεση της, ε, του πολιτισμού από τις συμφωνίες αυτές. Ο πολιτιστικός τομέας βοηθά στην ανάπτυξη της Ένωσης, αντιπροσωπεύει το 4,5% του ΑΕΠ και απασχολεί 8,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Θα επανέλθω σε αυτούς τους αριθμούς, γιατί πολλές φορές ακούμε διαφορετικά στατιστικά. Για μια στιγμή. Παρακαλώ να καθίσετε. So, Ces secteurs, disais-je, produisent du contenu. Παράγεται λοιπόν πολιτιστικό περιεχόμενο με καινοτόμες διαδικασίες που συναντούν την τεχνολογία με την τέχνη. Ο τομέας του πολιτισμού επιτρέπει επίσης και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή. Ανοίγονται νέες πρόπτικες το μέλλον της Ευρώπης επαφίεται στη νεότητά της, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης του τομέα αυτού είναι η σωστή λύση και θα βοηθήσει να επιστρέψουν οι νέοι στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των τομέων αυτών με άλλους οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός, να δούμε ακριβώς τις δυσκολίες που δημιουργεί το πέρασμα στον ψηφιακό κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαι πεπισμένη έχει να παίξει έναν πραγματικό ρόλο βοηθώντας να υπάρξει ένα σωστό διακανονιστικό πλαίσιο. Να υπενθυμίσουμε εδώ τη σημασία που έχουν προγράμματα όπως το Εράσμους για όλους και το Ευρώπη 2020. Η έκθεση που σας προτείνω ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της αγοράς, την αύξηση της εμβέλειας της αγοράς και την διατομεακή συνεργασία. Πέντε επιπλέον στοιχεία. Πρώτον θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας αξιόπιστες στατιστικές θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους του συγκεκριμένους τομείς, να ενισχύσουμε την παραγωγή την πολιτιστική με σωστές μορφές χρηματοδότησης, διευκόλυνση του περάσματος στον ψηφιακό κόσμο. Ας ξεκινήσουμε με τις στατιστικές. Σας έλεγα ότι οι στατιστικές που μας παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στο πρωινό ποικίλουν. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε έρευνες σε κάθε τομέα έτσι ώστε να έχουμε στοιχεία για την απασχόληση άμεση και έμεση στον τομέα αυτών των δραστηριοτήτων και τη σημασία και του βάρους τους στο ΑΕΠ των διαφόρων χωρών. Το να έχουμε αξιόπιστες και πρόσφατες στατιστικές είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει με επακριβέστατο τρόπο στις ανάγκες του τομέα. Παράλληλα, οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του τομέα αυτού μακροπρόθεσμα στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει μια ξεκάθαρη και διαρθρωμένη πολιτική γραμμή. Η πολιτική αυτή γραμμή θα πρέπει να συνοδεύεται και δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει σωστή επικοινωνιακή πολιτική. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην ισχυρή ικανότητα του πολιτιστικού τομέα να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Η ευαισθητοποίηση των νέων στον τομέα αυτό είναι καθοριστικό. Η εκπαίδευση στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού βοηθά επίσης και στην ισότητα των ευκαιριών και πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν αυτή τη μορφή στην εκπαίδευση. Η επαγγελματική κατάρτιση και η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τις σχολές και τις επιχειρήσεις είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ στις ανάγκες του τομέα αυτού. Να θυμίσω επίσης την σημασία που έχει να υποστηρίξουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση για τον πολιτισμό το ενωρίτερο δυνατόν και διαβίου. Τρίτον, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους τομείς αυτούς με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Η πρόεδρος είπε ότι προβλέπεται να υπάρξουν μειώσεις στον τομέα τον δημοσιονομικό. Εμείς θα πρέπει με νύχια και με δόντια να προσταθήσουμε να προστατεύσουμε τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Η χρηματοδότηση του τομέα είναι καθοριστική και θα πρέπει να αναζητήσουμε πολλαπλούς, ποικίλου, μικτούς τρόπους χρηματοδότησης μέσα σε ένα ελκυστικό και ευνοϊκό διακανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο, σαν παράδειγμα ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε επίσης τι ευκαιρίες ανοίγουν τα διαρθρωτικά ταμεία για την πολιτιστική παραγωγή και καλό τα κράτη-μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των πρωταγωνιστών του δημιουργικού τομέα στη χρηματοδότηση. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό που σας είπα το πέρασμα στον ψηφιακό κόσμο. Τον τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει κάποιες τεχνικές εξελίξεις πολύ σημαντικές προς την ψηφιοποίηση. Αυτή η αλλαγή δημιουργεί εμπορικές δυνατότητες αλλά παρουσιάζει και προκλήσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα σύγχρονο, ισορροπημένο, που να προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία και που να επιτρέπει στον καταναλωτή μια ποικίλη δυνατότητα πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο. Η παρουσία της παραγωγής μας στην διεθνή σκηνή είναι και αυτό κάτι που πρέπει να δούμε. Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πρέπει να θεωρείται δεδομένη στο διεθνές επίπεδο. Τώρα, πώς θα αγκυρώσουμε θα έλεγα την πολιτισμική παραγωγή με την τοπική οικονομία και κοινωνία. Οι προσπάθειες θα πρέπει πρώτα να γίνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και εδώ οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να καταστήσουν τις ίδιες τις περιφέρειες μοχλό για την ανάπτυξη. Κλείνοντας να πω ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας είναι το υπόδειγμα αυτού που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Εξαίρεση. Θα μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και η επιτυχία της προσπάθειάς μας θα εξαρτηθεί από την προσπάθεια ακριβώς που θα κάνουμε αλλά και από τα ταμεία και τις πιστώσεις τις οποίες θα έχουμε στη διάθεσή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Merci Marie-Thérèse. Je donne la parole à... Ευχαριστώ Marie-Thérèse. Ε, Ο Μπόρις έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Και σε αυτή την περίοδο μάλιστα που λαμβάνονται αποφάσεις για τον είναι σημαντική έκθεση. Τα κράτη-μέλη ετοιμάζονται για την ανανέωση των δημοσιονομικών προοπτικών Και είναι σημαντικότατο να υπογραμμίζεται στην έκθεση το βάρος, ε, το πόσο σημαντική είναι, σημαντικός είναι ο τομέας δημιουργικός για την οικονομία και την ανάπτυξη και δημιουργίες της απασχόλησης θα πρέπει να δίνονται, να τα χρήματα οι σωστές επενδύσεις από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Έχουμε και τον ορίζοντα 2020 που είναι ένα πρόγραμμα που προβλέπει την καινοτομία. Μπορούμε να έχουμε και καινοτομίε και στο δημιουργικό τομέα. Νέες τεχνολογικές λύσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον τομέα αυτό. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή και αρχίζουμε να μένουμε πίσω σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, επίσης διότι δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε τεχνολογικά. Η ΕΠΑ είναι πολύ πιο προχωρημένη σε αυτό και στο δημιουργικό τομέα. Πέρα από πιο πρακτικά ζητήματα όπως είναι η απλούστευση του φορολογικού συστήματος η καινοτομία θα μπορούσε να υποστηριχθεί και στο συγκεκριμένο τομέα που συζητούμε. Το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμπεριλαμβάνει πόρους για κατάρτιση σε διάφορους τομείς και ο τομέας που συζητούμε εμπίπτει στο στόχο οι άνθρωποι από τον τομέα αυτό, το καλλιτεχνικό, το δημιουργικό, θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένοι, να είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ε, ψηφιακής εποχής και τις ανάγκες της αγοράς. Τα τα ταμεία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, χορηγίες και δωρεές για επιχειρηματίες και όπως για εντελώς νέες επιχειρήσεις, για νέους, που ίσως θέλουν να αποφασίσουν να επενδύσουν χρόνο και οικονομικούς πόρους στον τομέα του πολιτισμού. Λοιπόν, χορηγίες, δάνεια, στον τομέα αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, να αναφέρω και τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο. Γνωρίζω αρκετά καλά το θέμα αυτό. Είναι πολύ δύσκολη η παρούσα κατάσταση. 70 με 80% των ευρωπαϊκών κινηματογράφων είναι ψηφιακοί, αλλά 20% των ευρωπαϊκών κινηματογράφων χρειάζονται ε, υποστήριξη για ένα-δύο χρόνια ακόμα, διαφορετικά θα κλείσουν. Και είναι πρόβλημα με κινηματογράφους που βρίσκονται σε μικρές πόλεις, κινηματογράφους που προβάλλουν κυρίως μη εμπορικές ε, ταινίες, Τώρα είναι η σωστή στιγμή λοιπόν να κάνουμε κάτι. Τελευταία φορά που θα μπορούσαμε να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα και να ψηφιοποιήσουμε όλους τους κινηματογράφους της Ευρώπης. Ε, συζητούμε την πρόσβαση εκατομμυρίων ανθρώπων στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, στις ταινίες, στον πολιτισμό. Άρα θα ήθελα Μαρή να υπογραμμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις τροπολογίες μου, ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών κινηματογράφων. Και αναφέρομαι και σε κινηματογράφους που έχουν οικονομικά προβλήματα που ίσως κλείσουν τον επόμενο χρόνο ή σε ένα-δύο χρόνια. Αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται, να τεθεί στο Συμβούλιο, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πέτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και τη Μαρή Τερέζ. Νομίζω πως ε, με την πρότασή σου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έθεσες ε, το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων για το μέλλον της δημιουργικής, ε, του δημιουργικού κλάδου στην Ευρώπη. Θα ήθελα να αφαιρθώ στη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Καταφέραμε να το τονίσουμε, το δέχτηκε η Επιτροπή από εμάς, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ακριβώς στον δημιουργικό αυτών κλάδων, να μην χαθούν όλα αυτά τα πράγματα κάπου στις επόμενες διαπραγματεύσεις για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί είναι κάτι το οποίο θεωρείται έτσι πάρα πολύ εύκολο να διαγραφεί και να γίνουν εκεί οι οικονομίες. πιστεύω πως πολλοί δεν το ήξεραν. Εγώ παραδείγματος χάρη χτες έμαθα πως 8% των εργαζομένων του Αμβούργου δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών, τον δημιουργικό και του πολιτισμού. Δηλαδή δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Κάτι το οποίο νομίζω μπορεί να συγκριθεί με τη βιομηχανική παραγωγή. Ένας δεύτερος τομέας ε, για τον οποίο λυπάμαι γιατί δεν είπε τίποτα η Κομισιόν αλλά εγώ θεωρώ πως είναι σημαντικό είναι η κοινωνική κατάσταση στον ε, τομέα αυτών. Εδώ πέρα μιλάμε για πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους, ε, ανασφάλιστους ή με συμβάσεις ε, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ε, έλλειψη κοινωνικής ασφάλειας που δεν δίνει σε πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους την δυνατότητα να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Είναι, ένα, εγώ θεωρώ, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν έφυξε η Κομισιόν. Όταν... Και πρέπει να το έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για αυτό τον κλάδο στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες πρέπει να επιζήσουν με ελάχιστα λεφτά και δεύτερον ε, τα κλασικά συστήματα ασφάλισης δεν μπορούν να τους ε, καλύψουν και στην περίπτωση της και στην περίπτωση χρεοκοπίας μιας εταιρείας Οπότε θα πρέπει νομίζω να το αναφέρουμε στην ε, έκθεση και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να κινητοποιηθούν και να φροντίσουν πως και οι απασχολούμενοι στον κλάδο αυτών να έχουν μια λογική κοινωνική ασφάλιση και να μην ε, κινδυνεύουν ανα πάσα στιγμή αν κάτι δεν πάει καλά. Αυτή δηλαδή η κοινωνική διάσταση πρέπει να μπει εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό το τομέα, δεν το έκανε δυστυχώς Κομισιόν και πρέπει νομίζω να το θίξουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μεγκάλσκι. Ευχαριστώ πολύ. Η Έμα Κλάρκ είναι σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους του ECR. Θέλω να παρουσιάσω τη δική της άποψη και εκ μέρους του ECR να πω και κάποια πράγματα αυτή η τομή είναι σημαντικότατη. Σημαντικότατη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Καλωσορίζει λοιπόν το ECR την αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια για το θέμα της ψηφιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης και της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Υποστηρίζουμε επίσης το θέμα το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, η προστασία των δικαιωμάτων αυτών είναι προαπαιτούμενο για την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Συμφωνούμε όλοι με την εισηγήτρια που αναφέρει ότι η περιφερειακή ανάπτυξη του τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η περιφερειακή και η τοπική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τομέα. Συμφωνούμε με την εισηγήτρια Τώρα, πιο αρνητικά στοιχεία. Θεωρούμε ότι κάτι λείπει ε, όσον αφορά την αναφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν μεγάλο κομμάτι του τομέα και παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Πρέπει να υπογραμμίσουμε λοιπόν τη σημασία τους διότι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να είναι ένας από, τις, ένας από τους βασικούς στόχους, προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πολιτισμού και του δημιουργικού τομέα. Νομίζω ότι είναι κρίσιμα σημεία που πρέπει να καλύπτονται στην έκθεση και ευχαριστώ την εισηγήτρια. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια. Νομίζω ότι εξηγεί πάρα πολύ, εξηγεί, συγγνώμη, πάρα πολύ καλά το διακύβευμα. Πράγματι ο κόσμος του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ε, είναι κάτι το ιδιαίτερα χρήσιμο. Συμβαίνει κάτι εδώ που συμβαίνει σε πάρα πολλά θέματα με τα οποία ασχολούμαι. Θα έχουμε πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες ανήκουν βασικά στα κράτη-μέλη. Και σε ορισμένα κράτη-μέλη πολλές φορές ανήκουν στις περιφέρειες και στις αυτόνομες περιοχές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες δράσης και μέσα στη διάθεσή της. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικά προβλήματα στον τομέα γενικότερα της χρηματοδότησης του πολιτισμού. Όταν μάλιστα υπάρχει μια οικονομική κρίση και υπάρχουν περικοπές, ο τομέας αυτός είναι ο πρώτος που πληρώνει την ύφη. Ο τομέας του πολιτισμού και ε, γενικότερα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε χώρες που όπως είπα οι αρμοδιότητες οι πολιτιστικές ανήκουν στα ίδια τα κράτη-μέλη. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Πράγματι, οι στατιστικές τις οποίες θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας για να βασίσουμε τη δράση μας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως αξιόπιστες, θα πρέπει να γνωρίζουμε το ποσοστό τη συγκεκριμένη αυτή οικονομική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ, θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσοι εργάζονται στον κόσμο του πολιτισμού. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία έτσι ώστε οι διάφορε κυβερνήσει που δεν τις απασχολεί πάρα πολύ ο τομέας του πολιτισμού θα πρέπει να ασχοληθούν έστω και σε οικονομικό επίπεδο γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ ισχυρή οικονομική δραστηριότητα. Τίθεται εδώ και το θέμα των διαφορετικών ταμείων, ένα πάρα πολύ σημαντικό <coughs> θέμα. Θα πρέπει να καλύψουν εν μέρη και τις ανάγκες του πολιτισμού και θα ήθελα να επιμείνω σε δύο επιπλέον θέματα. Το θέμα της Eh, Στο θέμα των χορηγών που θα πρέπει να το εξετάσουμε γενικότερα όχι μόνο στον τομέα του πολιτισμού, τα θέματα των ιδιωτικών χορηγιών αλλά και στα θέματα του αθλητισμού κτλ. Και εδώ υπάρχει θέμα για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές για να κατανοήσουν τα κράτη-μέλη τη σημασία αυτής της δραστηριότητας. Και δεύτερον θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη θα έλεγα φορολογική πολιτική σε σχέση με τα θέματα τα πολιτιστικά. Είναι καθοριστικό για τον κόσμο του πολιτισμού σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε επίσης και ο Σνάρφος Μουγκάλσκι για τα πνευματικά δικαιώματα. Εδώ τα πνευματικά δικαιώματα θα πρέπει να αναγνωριστούν πλήρως. Είναι πολύ σημαντικό για τους δημιουργούς και τα έργα τους και πάρα πολύ σημαντικό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί θυμίζω ότι η τεράστια πλειοψηφία των δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό γίνονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, Τόμας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την κυρία Σάντσε Σμιτ Πράγματι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια που έκανε. Ξεκινάμε από τρεις βασικές διαπιστώσεις. Πρώτον, την αναγνώριση της μεγάλης οικονομικής σημασίας του τομέα αυτού. Δεύτερον, η υποεκμετάλλευση σε εισαγωγικά του δυναμικού του συγκεκριμένου τομέα. Και τρίτον, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια διασύνδεση του τομέα αυτού με άλλα κομμάτια της οικονομικής δραστηριότητας και της τεχνολογίας. Κάτι το οποίο καθιστά τον συγκεκριμένο τομέα στρατηγικής σημασίας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να διαρθρώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την δημιουργικότητα και τον πολιτισμό με τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Εδώ να αναφερθώ σε κάποιες προτεραιότητες οι οποίες κατ' θα πρέπει να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν. Πρώτον, να υπάρξει γνωστοποίηση του σημαντικού δυναμικού του τομέα αυτού και των οικονομικών του δυνατοτήτων. Όπως το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, για να γίνει γνωστό το δυναμικό αυτό, θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστες στατιστικές στη διάθεσή μας. Ε, και δεν τις έχουμε ακόμα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια σωστή παρατήρηση του τομέα και κατά συνέπεια μια σωστή κατάρτιση ε, πληροφοριών γύρω από τον τομέα αυτό και στατιστικών στοιχείων. Οι αγορές πολλές φορές πράγματι στον τομέα του πολιτισμού είναι θα έλεγα εθνικές ή να το πω καλύτερα γλωσσικές και πολλές φορές η ευρωπαϊκή παραγωγή αντιμετωπίζει προβλήματα σε σχέση με τον παγκόσμιο χαρακτήρα της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Τρίτον, ε, το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε να κάνουμε με επιχειρήσεις οι οποίες ε, ε, είναι μικρές επιχειρήσεις και οι οποίες εκμεταλλεύονται το ταλέντο και τις δυνατότητες που έχει το ανθρώπινο δυναμικό τους. Ε, ένα επιπλέον θέμα είναι η σωστή κατάρτιση. Γνωρίζουμε ότι η κατάρτιση στον τομέα τον πολιτιστικό, ε, μερικές φορές και καλλιτεχνικό, έχει αρνητική εικόνα σε σχέση με το δυναμικό που παρουσιάζει η συγκεκριμένη παραγωγή. Όταν ένας ε, νέος, ένα παιδί λέει στους γονείς του θέλω να γίνω μουσικός ή θέλω να γίνω σχεδιαστής κινούμενων σκίτσων, ε, οι γονείς δεν λένε συνήθως ότι «Α, τι ωραία έχεις εξασφαλισμένο μέλλον παιδί μου». Λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε με πιο σωστό τρόπο την εικόνα αυτή. Και η εκπαίδευση επίσης ε, στον τομέα αυτό θα πρέπει να διασυνδεθεί καλύτερα με άλλους τομείς για τις ορισμένες χώρες η κατάρτιση των καλλιτεχνών παραμένει αρχαϊκού τύπου και δεν παραπέμπει στην χρήση νέων τεχνολογιών. Μια επιπλέον τέταρτη προτεραιότητα στα πλαίσια της ε, διασύνδεσης της παραγωγής της καλλιτεχνικής με άλλους τομείς υπάρχουν και οι κοινωνικές πλευρές. Μιλάμε για θέσεις απασχόλησης οι οποίες είναι πολύ προσωρινές. Κοινωνικά δημιουργούνται προβλήματα και θα έλεγα θα πρέπει εδώ ίσως να γίνουν προσπάθειες ενίσχυσης ενός αισθήματο ασφάλειας αυτών οι οποίοι ασχολούνται με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ένα επιπλέον θέμα είναι το θέμα της χρηματοδότησης ενός προγράμματος σε, ε, στην εναρκτήρια του φάση. Το βασικό πρόβλημα είναι να υπάρξει από την αρχή της δημιουργικής ε, διαδικασίας η κατάλληλη χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση πράγματι πρέπει να προέλθει από διαφορετικούς τομείς. Πρώτον, η αμοιβαία αναγνώριση με τους χρηματοδότες. Οι τράπεζες δεν είναι σε θέση ίσως στον τομέα αυτό με τις γνώσεις που έχουν να κάνουν καλά αυτή τη δουλειά και γι' αυτό δεν χρηματοδοτούν προγράμματα τα οποία είναι απολύτως βιώσιμα. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας δεν έχει την χρηματοδοτική ικανότητα που απαιτείται έτσι ώστε να είναι ελκυστικός. Ο τομέας αυτός έχει και κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που πολλές φορές τους αποκλείει από ορισμένε παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης Ξέρουμε ότι έχει σαν παράδειγμα πολύ μικρό εργατικό δυναμικό και αυτό πολλές φορές λειτουργεί αρνητικά. Ε, πάντως μέσω των μηχανισμών εγγυήσεων των δανειοδοτήσεων κάποιες λύσεις θα πρέπει να βρεθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να θέσει στη διάθεση του τομέα τα απαιτούμενα μέσα. Θα πρέπει φυσικά να μην θεωρούνται τα προϊόντα που παράγει ο τομέας αυτός απλά εμπορικά προϊόντα. Υπάρχει και άλλη μία πλευρά και άλλη μία προτεραιότητα. Εδώ το δημόσιο, οι δημόσιες αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο, ε, πιο διαφορετικό θα έλεγα από άλλους τομείς. Καταρχάς ρυθμίζουν σε επίπεδο διακανονιστικό και φορολογικό την παραγωγή αυτή και κυρίως διευκολύνουν συνοδευτικά την πολιτιστική και καλλιτεχνική παραγωγή και έχουν πολλές φορές οι δημόσιες αρχές και το ρόλο του παραγωγού τέτοιου είδους πολιτιστικών προϊόντων. Κάποιες αγορές τέτοιες, κάποιες δραστηριότητες καλλιτεχνικές, πνευματικές, πολιτιστικές από τη φύση τους δεν μπορεί να είναι προσοδοφόρες οικονομικά, αλλά είναι απαραίτητες και χρήσιμες και εκεί τίθεται το θέμα της χρησιμότητας του δημόσιου τομέα, της κρατικής παρέμβασης. Και εδώ θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τομεί αυτοί λοιπόν μέσω των νέων τεχνολογιών αντιμετωπίζουν νέες μορφές προκλήσεων. Δεν θα πρέπει τις εξελίξεις αυτές να τις γιατί έτσι θα καταδικάσουμε την καλλιτεχνική και πνευματική παραγωγή. Ο ανταγωνισμός παγκοσμίω είναι ισχυρότατος και πρέπει επίσης να τεθεί και το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια γιατί επιμένει και στον σημαντικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και στην αγκύρωση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας στο τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Οι τοπικοί παράγοντες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την προστασία τέτοιων δραστηριοτήτων, για την ανείχνευση και προώθηση νέων ταλέντων και πρέπει να υπάρξει μία θα έλεγα τοπική και περιφερειακή μορφή διαχείρισης της πολιτιστικής παραγωγής. Ευχαριστούμε. Τον λόγο έχει η Κομισιόν. Mm. Η κυρία Τωρότα Νίγκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το κείμενό της. Καλωσορίζουμε την, ε, το κείμενο και σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι διάφορα σημαντικά στοιχεία της ανακοίνωσής μας έχουν ληφθεί υπόψη. Αυτά που υπογραμμίστηκαν περισσότερο ήταν το θέμα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και οι προκλήσεις της ψηφιακής παγκοσμιοποίησης και η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και η περιφερειακή ανάπτυξη, ξεκινώ με μια διευκρίνηση. Το σημείο για το Horizon και το πεδίο εφαρμογή για το στόχο και το πεδίο εφαρμογή ανακοινώσεως. Ε, πρέπει να μην υπάρξουν παρανοήσεις. Η ανακοίνωση λοιπόν του Σεπτεμβρίου 2012 καθορίζει μια στρατηγική με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Η βραχυπρόθεσμη φιλοδοξία σχετίζεται με ομάδα δράσεων που θα εφαρμοστούν συντονισμένα και από διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά από την υιοθέτηση της ανακοινώσεως πάνω από 60 διαφορετικές δράσεις επί πέντε αξώνων πολιτικής έχουν εφαρμοστεί. Και είμαστε πεπισμένοι ότι έτσι ενισχύεται ο συντονισμός των μέσων και αυτό θα είναι εφικτό και εντό των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών. Έχουμε βέβαια και μακροπρόθεσμους στόχους της στρατηγικής. Θέλουμε ο πολιτισμός και ο δημιουργικός τομέας να είναι στο επίκεντρο του, της στρατηγικής Ευρώπης για το 2020. Και ανακοίνωση καλεί τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν πολυεπίπεδες στρατηγικές για να προωθήσουν το δυναμικό της δημιουργικότητας καινοτομίας στον τομέα του πολιτισμού και να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο στα αναπτυξιακά σχέδια τα εθνικά. Μιλάμε για εθνικά αναπτυξιακά σχέδια και στρατηγικές. Και για μας αυτή είναι, αυτός είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον τομέα του πολιτισμού. Και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει στενή σχέση, ρεαλιστική, με τη νέα πολιτική συνοχής και τον στατηγικό προγραμματισμό για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Σημειώνουμε το αίτημα να δημιουργηθεί ένα φόρουμ των εμπλεκομένων φορέων για τον τομέα που συζητούμε. Το πρόγραμμα εργασιών για τον πολιτισμό 2011-2014 θέτει το διάλογο με τους εμπλεκομένους φορείς σε ύψιστο επίπεδο και απαιτεί και συντονισμό. Είναι βασικά εργαλεία για τη δράση Ευρωπαϊκής Ενώσης στον τομέα του πολιτισμού. Η πλατφόρμα για την ανάπτυξη του δυναμικού του τομέα δημιουργήθηκε το 2008. Πάνω από 40 οργανισμοί συμμετέχουν στην προσπάθεια, εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα του δημιουργικού τομέα ε, και έχουν κάνει διάφορες προτάσεις και θα εξακολουθούν να είναι ενεργοί. Ο διαθρωμένος διάλογος όμως με αυτούς τους εμπλεκομένους φορείς και η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού αξιολογούνται. Ανάλογα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης, ίσως εξετάσουμε ενδεχόμενη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως προβλέπετε και στο σχέδιο κειμένου. Όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, προτιμούμε να αναφερόμαστε σε πρόσβαση στη χρηματοδότηση και όχι χρηματοδότηση αυτή αυτή. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε συμπληρωματικότητα του μηχανισμού της οικονομικής στήριξης με το CCS. Προφανώς έχουμε δύο μέσα Έχουμε τα μέσα εγγύησης που αναφέρθηκαν, που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ιδιωτική χρηματοδότηση, γνωρίζοντας τα προβλήματα όσον αφορά τα άειλα στοιχεία ενεργητικού για τις επιχειρήσεις του τομέα και έχουμε τη δυνατότητα για τη δημιουργική Ευρώπη της ανιοδότησης αλλά και στο πρόγραμμα κόσμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επανειλημμένα αναφέρθηκαν αυτές σήμερα και το μέσο που προβλέπεται στο Horizon 2020. Έχουμε, θα έχουμε χορηγίες συγκεκριμένες για τη στήριξη της ευρωπαϊκής διάστασης, για την καινοτομία, για το επιχειρηματικό πνεύμα στον τομέα. Σημειώνουμε όντως την αναφορά του, της μικτής χρηματοδοτήσεως. Είναι σημαντικότατο στοιχείο. Όμως, η στήριξη προ τι επιχειρήσει αυτέ δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο πλευρά οικονομική στήριξη. Αυτό είναι ρόλο των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να δημιουργήσουν τι κατάλληλε συνθήκε για τη βιομηχανία του, του δημιουργικού αυτού τομέα, πέρα τη χρηματοδότηση. Άρα χρειάζεται και το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο. Πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε επανειλημμένα. Και το κείμενο δίνει πολύ καλά παραδείγματα αυτή τη προσέγγιση. Όσον αφορά λοιπόν το IPR, ξέρετε, ότι γίνεται διαβούλευση με τους εμπλεκομένους φορείς και ονομάζεται Licenses for Europe και όπως αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας, η διαδικασία αναθεωρήσεως του νομικού πλαισίου για τον τομέα το δημιουργικό θα λάβει χώρα. Διεθνείς τύχε. Ακροθυγώς να αναφερθώ στον ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και την ομάδα που συζητά εξαγωγικέ στρατηγικέ για το δημιουργικό τομέα. Η ομάδα ετοιμάζει ένα χειρίδιο καλών πρακτικών. Βλέπει ποια είναι τα καλά παραδείγματα που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τι εξαγωγέ πολιτισμικών προϊόντων. Και αυτό για όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι πολύ σημαντικό. Να έχουμε μια εικόνα. Να μάθουμε ένα από τον άλλον. Να αντισταθούμε στι πιέσει από χώρε όπω είναι η Κίνα. Η Νότια, Κορέα, η Ινδία, που παράγουν πολλά στο δημιουργικό τομέα. Τέλος. Θέμα ιδιαίτερο σημαντικό για μας. Διατομιακή καλλιέργεια διαφόρων τομέων πολιτικής δημόσιας και πώς ο πολιτισμικός τομέας επηρεάζει τη δημόσια ζωή εν γέννη. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και αποτελέσματα υπερχείλησης από τομέα σε τομέα δηλαδή του πολιτισμικού τομέα σε άλλους τομείς πολιτικής. Το ανέφεραν διάφοροι. Μπορεί αυτό να αναφέρεται εκτενέστερα στην έκθεση. Να φαίνεται πως οι τομείς της δημόσιας ζωής επηρεάζονται από το πολιτισμικό. σημαντικό ταμεία. τάτο. Τώρα είναι η στιγμή σωστή που ετοιμάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα διευθυντικά ταμεία, τα κράτη-μέλη. Πιστεύουμε ότι είναι σωστή προσέγγιση. χρειάζεται επενδύσεις στον πολιτισμικό τομέα και δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από τα στρατηγικά προγράμματα επενδύσεις. Γι' αυτό καλωσορίζουμε το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που ετοιμάστηκε στην Επιτροπή Ρέτζι, που ασχολήθηκε με το θέμα. Ευχαριστώ εκ νέου την εισηγήτρια. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενημερωτικά τα όσα μας είπατε. Και ευχαριστώ ιδιαίτερο την κυρία για όσα μας είπε. Μας έδωσε μια άποψη εκ των έσω των τεκτενωμένων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάνατε μετά την ε, χειμερινή σας σύσταση. Πολύ καλά αυτά που μας είπατε. Έπρεπε να σας το πω. Κύριε Μιγκάλσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, λέει ο Μιγκάλσκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σύντομα έχω ένα σχόλιο. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπατε όσον αφορά τα όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω κάτι όμως. Σε δημόσιες α, δηλώσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να αποφεύγετε να αναφέρετε ότι η Κίνα είναι το μοντέλο μας, το παράδειγμά μας, κυρίως όσον αφορά τον πολιτισμό. Συμφωνώ ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε τα επιτεύγματα, τα οικονομικά της εν λόγω χώρας. Όμως δεν είναι δημοκρατική χώρα. Πόρα απέχει από την ορθή αντιμετώπιση των πολιτών της. Αυτή είναι η χώρα που είναι πολύ καταπιεστική, που παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών της. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Θα πρέπει να το θυμόσαστε αυτό όταν μιλάτε δημοσία. Κατηδίαν μπορούμε να κουβεντιάσουμε την Κίνα με διαφορετικό τρόπο. Σας προειδοποιώ όμως μην κάνετε τέτοιου είδου ε, αναφορές όταν μιλάτε για την Κίνα. Ευχαριστώ. Ναι, σας παρακαλώ. Κύριε Μιγκάλσκι, το θέμα δεν αφορά τώρα το πολιτικό σύστημα. Μπορεί να συμφωνούμε μαζί σας. Ε, πράγματι Βλέπουμε τι κάνει η Κίνα και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Τώρα, ακούγοντα την Κομισιόν, βεβαίω τόνισε πω ε, και τα διαρθρωτικά ταμεία παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Αυτό, ναι, πάντα έτσι ήταν, αλλά δυστυχώ βλέπουμε εδώ πέρα στι προτάσει των διαρθρωτικών ταμείων δεν υπάρχει καν η λέξη πολιτισμό εκεί μέσα και πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό το οποίο είπατε δηλαδή κάπου πρέπει να το δει η Κομισιόν να μπει ο πολιτισμός κάπου στα, στα διαρθρωτικά ταμεία. Και το έχουν πει και άλλοι νομίζω και στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων κτλ. Υπάρχει κάποιο άλλο, Μαρή Τερέζ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ευχαριστώ τους συναδέλφους για όλες τις προτάσεις τους. Ακριβέστατες ήταν. Ντόρις δίκιο έχεις. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκανε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και έδωσε ενδείξεις. Προβληματίζομαι όλος ιδιαίτερος όσον αφορά τη δυνατότητά μας να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα που να μπορούν να εφαρμοστούν και που να έχουν πραγματικά αποτελέσματα. Όσον αφορά τα θετικά ταμεία, Πραγματική σημασία έχουν, τα αναφέρω τακτικότατα τα ταμεία αυτά και πολεμώ τους ώστε να χρησιμοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού. Είμαι μέλο τη Επιτροπή Ρέτζη και κατέθεσα τροπολογίε όσον αφορά τον κανονισμό των ιδιωτικών ταμείων, ώστε ο πολιτισμό να λαμβάνεται υπόψη. Ακόμα γίνεται διάλογο, ε, τριμερή διάλογο, αλλά με υποστηρίζουν πάρα πολλά μέλη τη Επιτροπή μου, ε, Επιτροπής μου ανεξάρτητα από την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουν. Στην κυρία Καμεβέρτη και σε εκείνου που ανέφεραν τη σημασία των Εθνικών Ταμείων έχω να πω αυτό. Υπάρχει μια πραγματική δυνατότητα και λόγω της οικονομικής σημασίας πάνω από 300 δις τα διαθωτικά ταμεία μπορούν πράγματι να δώσουν βοήθεια επιτόπου και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς αυτό το σκοπό. Εξάλλου επανειλημμένα αναφέθηκε σημαντικός ρόλος του δημιουργικού τομέα για την οικονομία και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να πείσουμε λοιπόν τους ερετούς ε, εκπροσώπους που χρησιμοποιούν τα επιχειρησιακά προγράμματα ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πολιτισμός. Όχι μόνο σαν αντικείμενο ή περιθωριακό θέμα που αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, συμμετέχει πράγματι στην οικονομία και την ανάπτυξη ο δημιουργικό τομέας. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Πρέπει να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε. εκείνοι που χρησιμοποιούν τα προγράμματα ειδικού τομέα μας ζητούν να δραστηριοποιηθούμε για να χρησιμοποιηθεί το ΜΑΣ. Αναφέρθηκαν ανησυχίες όσον αφορά την κατάρτιση. Ε, είναι αρμοδιότητά μας. Θα πρέπει να προτείνουμε μέτρα που θα δώσουν κίνητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι έχει ληφθεί υπόψη αυτή η πτυχή. Και η Σαμπέλ Τωμά το ανέφερε. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε πραγματικά την επαγγελματική κατάρτιση, την εναλλακτική προσέγγιση. Στις περισσότερες χώρες δεν χρησιμοποιείται επαρκώς. Θεωρείται σαν ένας χώρος στάθμευσης, αν θέλετε, δευτερευούση σημασία σε σχέση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά δίνει υπεραξία η κατάρτιση στον οικονομικό τομέα. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες ενημέρωσης και επικοινωνίας πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με αυτούς τους τομείς. Υπάρχουν δομέ για και θα πρέπει να γνωστοποιηθούν. Σημείωσα τις ε, ανησυχίες όσον αφορά τη σημασία που πρέπει να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικονομικά, να δώσουμε σημασία, είναι πάρα πολύ σημαντικές πράγματι, εκπροσωπούν πάρα πολλές τις απασχόλησης, κυρίως μέσω υπεργολαβιών, μπορούμε με επιδοτήσεις να χρηματοδοτήσουμε άμεσα, αλλά και με συνοδευτικά μέτρα έμεσα μέσω τραπεζών, μέσω μηχανικής στήριξης ε, και να υπάρχει μεικτή χρηματοδότηση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χρηματοδότηση. Υπάρχει και μέσος τρόπος συμμετοχή στη χρηματοδότηση. Μέσω της φορολόγησης θα πρέπει να δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις όσον αφορά τα πολιτισμικά αγαθά. Όσον αφορά την υποεκμετάλλευση ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι, να προβάλλουμε το δημιουργικό και πολιτισμικό τομέα περισσότερο. Όλοι γνωρίζουν ότι τα πολιτισμικά αγαθά και τα δημιουργικά αγαθά δεν είναι απλά εμπορεύματα όπως τα άλλα και έτσι πρέπει να τα προβάλλουμε. Σημείωσα αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους μακροπρόθεσμους στόχους. Πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πραγματικές στρατηγικές για τον πολιτισμικό τομέα. Και ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται μια πραγματική βάση δεδομένων, στοιχεία, για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον τομέα. Να του δώσουμε μεγαλύτερη ορατότητα. Περιμένω να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις έμεσες συνέπειες που έχει ο τομέας για άλλους τομείς της κοινωνίας. Ο δημιουργικός και πολιτισμικός τομέας ε, μπορεί να βοηθήσει στην ε, κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση. και να προωθήσει τομείς πέρα της παιδείας. Το τελευταίο που έθιξε ο κ. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κίνα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σημασία της Κίνας στον τομέα τα οικονομικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, την παραποίηση, την αντιγραφή. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει παραποίηση και αντιγραφή τομέα. Είναι πάρα πολύ ε, ε, στην εντυπωσιακή οικονομική σημασία που έχει το τομέας. Χρειάζονται μέτρα για την προάσπιση της πνευματικής ιδιοκτησίας και εκεί μπορούμε να παρέμβουμε. Χθες ο Μισελ Μπαρνιέ μίλησε στην Ειδική Επιτροπή ΚΡΙΜ και αναφέρθηκε στον τομέα. Το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ληφθούν όμως συγκεκριμένα μέτρα προστασίας ε, του τομέα. Ευχαριστώ Μαρή Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως κάποια από αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ πέρα στο νέο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη έχουν ε, υποβληθεί και γραπτό στο θέμα μιας τράπεζας δεδομένων. Πιευτόμαστε αν μπορούμε να το εμπιστευτούμε στο οπτικό ακουστικό παρατηρητήριο. Πρέπει να ξεκαθαριστεί εμπάσφερτος και με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά δεν γίνεται χωρίς να συνεννοηθούμε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και πρέπει να δούμε αν έχουν τα εφόδια για κάτι τέτοιο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερον, η... ο δημιουργικό κλάδο, όπω είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μα είπατε για το Αμβούργο, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και στην Κολονία και στο Μόναχο. Εκεί πέρα είναι τρεις ε, μεγάλες εστίες ε, πολιτισμού και κινηματογράφου. Δεν είναι το Βερολίνο. Το θέμα βέως είναι πάντα το ότι αν δεν λύσουμε το ζήτημα του copyright τότε ε, χάνεται το οποιοδήποτε πλέον έκτημα. Οπότε η έκθεση αυτή Δεν περιέχει επίσης την, τις λέξεις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Θα ήθελα τουλάχιστον κάπου να αναφερθούν. Η σκέψη υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει η λέξη. Η δημιουργική Ευρώπη την έχουμε αναφέρει ρητός. Νομίζω μπορούμε να αναφέρουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα Μέχρι την 5η 12 η ώρα πρέπει να έχουμε έτοιμες τροπολογίες. Αυτό προβλέπουν οι κανόνες. Του χρόνου λίγη εντολή μας, γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε κάπως πιο γρήγορα. Μέχρι την 5η στις 12, λοιπόν, μεθαύριο, πρέπει να έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες, αλλά νομίζω πως τα έχετε όλοι σε όλες τις γλώσσες, οπότε δεν θεωρώ πως είναι πρόβλημα και τα υπόλοιπα νομίζω τα κάλυψε όλα η Μαρή Τερέζ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία 2010-2012. Ο κύριος ε, Γεωργιος Παπα-Νικολάου ε, νομίζω θα μας εξηγήσει τα σχετικά. Παρακαλώ. Ε, Thank you, Madam Chairwoman. This report comes in response to the Commission. Αυτή η έκθεση ανταποκρίνεται στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, strategy for Youth. If you remember, we had ε, an introduction in the... Είχε υπάρξει μια εισαγωγή λοιπόν γύρω από τις μελέτες αυτές πριν μερικά χρόνια. Τώρα φτάνουμε στο τέλος του πρώτου κύκλου και θα πρέπει να αναφερθούμε στα βήματα πρόοδου που έχουν γίνει. Η έκθεση αυτή έρχεται τώρα με μια κάποια καθυστέρηση. Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων έγινε στην Επιτροπή μας το προηγούμενο φθινόπορο. Υπήρξε μια διαφορά με την Επιτροπή Απασχόληση σχετικά με τα άρθρα που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν η Επιτροπή Απασχόλησης δυστυχώς είναι η, αρμόδια επί της Είχαμε πολύ περιορισμένο χρόνο και για τις μεταφράσεις. Ελπίζω πάντως ότι όλοι οι συνάδελφοι θα κατανοήσουν το βιαστικό του πράγματος. Οι προκλήσεις των νέων είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισε το Συμβούλιο να κάνει μια συνάντηση κορυφής μόνο για τα θέματα της νεότητας, των νέων. Η κατάσταση είναι προβληματική και στον τομέα της απασχόλησης και στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα της έλλειψης συμμετοχής ε, που παρατηρείται Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις της έκθεσης μας. Έχουμε προχωρήσει στον καθορισμό τριών κύκλων εργασίας, όπως σας προανέφερα. Εμείς προσπαθήσαμε να δούμε τι πετύχαμε μέχρι τώρα και τι όχι και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτή την προσπάθεια. Ε, πράγματι η πρόοδος έχει υπάρξει σε κάποιους τομείς, αλλά η κρίση που βιώνουμε επηρεάζει πάρα πολύ πολλούς από τους νέους και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε προτεραιότητες, να ιεραρχήσουμε τα πράγματα, να δούμε τι είναι επίγον και να ξεκαθαρίσουμε τον ορίζοντα. Ήδη έχουμε λάβει υπόψη τις νέο της Επιτροπής Απασχόλησης, Λάβαμε επίσης υπόψη και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νεότητα το 2012 και τις δραστηριότητες των υπολείπων επιτροπών για το πρόγραμμα ΓΕΣ, για το πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ και επίσης την έκθεση της συναδέλφου Ντεβεντάλοβα. Εμείς προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να προβλέψουμε για τον επόμενο κύκλο της στρατηγικής για τους νέους. Όπως σας είπα πριν, αυτό το οποίο επιλέξαμε εδώ είναι να υπογραμμίσουμε κάποια κεντρικά θέματα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χώρο θα έλεγα, η έκθεση δεν εξαντλεί όλους τους τομείς. Ε, το κείμενο όπως είπα δεν μπορεί να γενικεύει λόγω της κρίσης αλλά πρέπει να ιεραρχεί με απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Περιγράφουμε την σημερινή κατάσταση, προσπαθούμε να συνδυαστούμε με τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στην Επιτροπή μας και με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές έτσι ώστε στο μέλλον να υπάρξει ένας οδικός χάρτης ο οποίος να είναι χρήσιμος στην Επιτροπή για το μέλλον. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για τα επίπεδα ζωής των νέων στην Ευρώπη σήμερα. Αυτό το έχουμε συζητήσει. Στον τομέα της παιδείας, λόγω της κρίσης, πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε περικοπές. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι περικοπές αυτές ξεπερνούν το 10% και αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη γιατί πράγματι βλάπτει ό,τι έχουμε πετύχει στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Απαιτούνται περισσότερα μέσα χρηματοδότησης από ό,τι στο παρελθόν και επίσης ε, προώθηση προγραμμάτων όπως το Εράσμος για όλους. Έτσι θα είναι ο σωστός δρόμος. Ο εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης είναι μια μεγάλη θα έλεγα πρόκληση για την Ευρώπη. Ε, ο καλύτερος τρόπος για να προωθηθεί η καινοτομία είναι η παιδεία και δεν αναφέρουμε μόνο στην επίσημη παιδεία. Παρατηρούμε να υπάρχει μια έλλειψη αποτελεσματικότητας σε διάφορες χώρες για την αναγνώριση της μη τυπικής θα έλεγα ε, εκπαίδευσης θα πρέπει να προωθήσουμε την κριτική σκέψη ε, και την εφευρετικότητα. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, λειτουργούν δύσκολα γιατί αλλάζουν συνεχώς. Οι νέοι που είναι εκτός ε, απασχόλησης και παιδείας εξεπερνούν το 23% ένα στους 4. Αυτά είναι απαράδεκτα και πρέπει να αντιμετωπιστούν γενικά σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανεργία ανάμεσα στους νέους έχει αυξηθεί, φτάνουμε στο 55, 60, 65% απαράδεκτα επίπεδα. Είναι προκλητικό ταυτόχρονα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να μην χρησιμοποιούνται στα διαφθορτικά ταμεία, ιδιαίτερα στο κοινωνικό ταμείο πρέπει να δοθεί ε, θα έλεγα προσοχή στην καλύτερη χρηματοδότηση μέσω των ε, περιφερειακών, των διαφορετικών συγγνώμη ταμείων. Ε, θα πρέπει επίσης να εφεύρουμε και διαφορετικά μέσα στήριξης της εφευρετικότητας και της καινοτομίας. Η task force ε, για τους νέους δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες αλλά δεν έχουμε πάρει ακόμα εκθέσεις δραστηριότητας και ελέγχου της δραστηριότητας αυτής. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερες προσπάθειες. Έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο επίσης για τη συμμετοχή των νέων, όχι γιατί αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά γιατί τα περιθώρια για την εμπλοκή των νέων είναι πάντα αρκετά μεγάλα. Όπως είπα στην αρχή της παρουσίασής μου προσπαθήσαμε να επιμείνουμε σε κάποιες προτεραιότητες. Νομίζω ότι πάντα οι νέοι θα πρέπει να είναι συνεχώς online, θα πρέπει να έχουν ε, μέσα ε, στη διάθεσή τους Πρέπει να τους βοηθήσουμε να το πετύχουμε αυτό, να τους ακούσουμε και να δράσουμε μαζί τους στο διαδίκτυο γιατί εκεί είναι οι νέοι. Θα πρέπει να προσέξουμε τι θέλουν για να καθορίσουμε τις πολιτικές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθοδηγήσει τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα από ό,τι τώρα στον επόμενο κύκλο της στρατηγικής. Δεν αρκεί συνάδελφοι να πούμε ότι έχουμε τα κατάλληλα μέσα όπως το ανοιχτή μέθοδο συντονισμού και απλά εφαρμόζουμε τα μέσα αυτά. Όχι, απαιτούνται περισσότερα. Ένα τέτοιο κείμενο είναι δυναμικό από τη φύση του, προσαρμόσιμο και ζητάμε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε τα κράτη-μέλη στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου να λάβουν υπόψη τους τις εκθέσεις μας, εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα σας απασχολήσω άλλο. Νομίζω ότι τη συζήτηση αυτή μπορούμε να τη συνεχίσουμε για πάρα πολλές ώρες, θα συνεχιστεί για πολλούς μήνες έτσι κι αλλιώς και νομίζω θα συνεχίσουμε τις ανταλλαγές ε, απόψεων με τους συναδέλφους. Ε, όσοι επιθυμούν μια πιο προχωρημένη ανάλυση μπορεί να διαβάσουν την αιτιολογική έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις, Ντεβεντάλοβα, Ταβάρες, Μακάλκιν, Βερζιά, γιατί πράγματι έχουν προσφέρει πολλά στις συναντήσεις που είχαμε μαζί τους. Πολλές από τις ιδέες τους προσπάθησα να ενσωματώσω στο κείμενο. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Λεζέν, τον διευθυντή της αρμόδιας διεύθυνσης, για την αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει. Είναι μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και κυρίως την κυρία Φάμπια Φοντανέλη για την υπομονή της. Νομίζω ότι με την έκθεση αυτή κάτι μπορούμε να προσφέρουμε σημαντικό και σίγουρα και οι τροπολογίες των συναδέλφων θα είναι χρήσιμες, πολύτιμες και θα προσπαθήσουμε να τις εντάξουμε στο κείμενο. Ας προσπαθήσουμε να δείξουμε για μια ακόμη φορά την αποφασιστικότητά μας να βοηθήσουμε τους νέους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιγκάλσκι έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο εισηγητής μας ανέφερε πως είχε την ευχαρίστηση να συνεργαστεί με την κυρία Μακλάρκιν. Οπότε θα ε, επικοινωνήσετε και μαζί μου και ελπίζω και η δική μας συνεργασία να είναι ικανοποιητική. Λίγα λόγια λοιπόν για την έκθεση αυτή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι με το σχέδιο αυτό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε τις σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Σημαντικό αυτό. Επίσης υποστηρίζουμε το ότι η έκθεση το σχέδιο έκθεση ορίζει τα του προγράμματος ε, για τον πολιτισμό και την θετική, ε, το θετικό αντίκτυπο που έχει η έρευνα και η ανάπτυξη στις, ε, στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα της δημιουργίας νέων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως ε, ευρωπαϊκές σπουδές στα προγράμματα των πανεπιστημίων. Αυτό κατά την άποψή μας δεν είναι δεν ανήκει στο αντικείμενο της έκθεσης αυτής και δεν είναι αναγκαίο. Επίσης καλωσορίζουμε το ότι η έκθεση αυτή δίνει μεγαλύτερο βάρος στη σημασία του αθλητισμού και της ε, άθλησης ε, και η κυρία Μακλάρκιν ε, υπογραμμίζει και τονίζει πως νους υγιής εν σώμα τη Γη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει και για το ότι έλαβε υπόψη τις συστάσεις και τα σχόλια των σχεδόν συγκητών. Συμφωνώ μαζί του πως είναι απογοητευτικό πως σε κάποια κράτη-μέλη έχει γίνει πάρα πολύ λίγη μικρή πρόοδος και σε κάποιες περιπτώσεις έχει επιδεινωθεί η κατάσταση για τους νέους ανθρώπους. Είναι σαφές πως με το έγγραφο αυτό πρέπει ξεκάθαρα και με ουσιαστικό τρόπο να αναφέρουμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους, τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις όμως θεωρώ πως είναι επίσης αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Ενώ ζητήματα όπως η ενέργεια των νέων και αυτών οι οποίοι δεν βρίσκονται σε κάποια κατάρτιση και εκπαίδευση είναι γνωστά ε, καλωσορίζω το ότι αναφέρεται το τι περαιτέρω επιπτώσεις έχουν αυτά τα φαινόμενα και τα ζητήματα επίσης πνευματικής υγείας. Υπάρχει λοιπόν επίσης ε, το ζήτημα της ε, χρηματοδότησης ε, των προγραμμάτων αυτών. Αλλιώς, στα κρατημέλη αλλιώ δεν θα είναι ποτέ αποτελεσματικά τα προγράμματα. Αυτά εκπαίδευση και κατάρτισης κάπως αντιμετωπίζουν το άμεσο πρόβλημα, αλλά τα παράγωγα προβλήματα, δηλαδή το ότι οι νέοι αναγκάζονται να δουλεύουν σε προσωρινές δουλειές που δεν έχουν σχέση με την ειδίκευσή τους και χωρίς μακροπρο... μακροχρόνιες προοπτικές, ε, είναι εξίσου σοβαρά. Επιπλέον τα προβλήματα δεν θα περιοριστούν μόνο σε αυτή την γενιά, αλλά οι μελέτες δείχνουν πως όσοι ξεκινάνε τη σταδιοδρομία τους υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αβεβαιότητα, ε, πιθανότατα θα έχουν και άλλες περιόδους ε, αβεβαιότητας και ανεργίας στο μέλλον και ε, καθώς υπάρχει ακριβώς η έλλειψη αυτοπεποίθησης νωρίς στην ζωή τους. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η ρητορική της στιγμής μιλάμε είναι για μια χαμένη γενιά, χωρίς ευκαιρίες, χωρίς ελπίδα και χωρίς μέλλον. Όμως, όταν συναντάει και βλέπει κανείς τους νέους, είναι σαφές πως κανένας νέος δεν θέλει να κατηγοριοποιηθεί έτσι και να περιμένει να περάσει η οικονομική κρίση. Εγώ καλωσορίζω τη θέση του εισηγητή και θεωρώ πως εδώ πέρα υπάρχει μια σοβαρή βάση για μια σωστή στρατηγική για τους Ευρωπαίους νέους και καθώς προχωράει η συζήτηση βεβαίως θα υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες που ελπίζω να βοηθήσουν την ε, έκθεση και αναμένω και τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βινταλόβα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εν πρώτης εκτιμώ την έκθεση που υπευλήθη από τον κύριο Είναι μια πολύ καλή, ισορροπημένη έκθεση και τα επιχειρήματά του είναι τα ίδια αυτά που συνήθως εκφράζονται στην Επιτροπή μας. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που μας είπε, διότι μίλησε ε, με πολύ συνετό και σοφό τρόπο και συμφωνώ μαζί του πρέπει να τονίσω ότι έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη στρατηγική για τους νέους. Η αρχή της επικουρικότητας υπάρχει και σε κάποιο βαθμό δεσμεύει, μας δένει τα χέρια αυτή η αρχή. Ελπίζω όμως ότι η στρατηγική για τους νέους ως παρουσιάζεται τώρα θα αποτελέσει τροφή προσκέψη αυτό που εκτιμώ και που αναφέρεται στην έκθεση είναι η πτυχή των νέων τεχνολογιών, πώς μπορούμε να επικοινωνούμε με τους νέους, πώς μπορούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω οι νέοι. Δεν αρκεί να αναφέρουμε όλα τα προβλήματα και μόνο που αντιμετωπίζουν οι νέοι, πρέπει να αναφέρουμε και είναι σημαντικό αυτό να προτείνουμε και κάποιες ε, λύσεις και διεξόδους. Οι οργανώσεις των νέων, παραδείγματο χάρη, έχουν πολλά περιθώρια ελιγμών, Μεγάλα περιθώρια. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε οι οργανώσεις των νέων ε, τι ακριβώς μας λένε. Οι νέες τεχνολογίες που αναφέρονται στην ε, έκθεση είναι ένας τομέας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία, να χρησιμοποιηθεί για να παράσχει νέες δεξιότητες στους νέους. Δεξιότητες που θα μπορούσαν οι νέοι να χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους και αυτό σχετίζεται στενά με τη μεταρρύθμιση του τομέα της παιδείας και θα υποβάλω σύντομα κάποιες προτάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν πολλοί νέοι που είναι άνεργοι και οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση η οποία έχει ζήτηση στην αγορά. Σχετικά με αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θα ήταν καλό να αναγνωρίζεται και η άτυπη ε, εκπαίδευση. Και ελπίζω οι εθελοντικές δραστηριότητε να εξακολουθούν να υποστηρίζονται από, τις, ε, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εν γέννη είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που παρουσιάστηκαν, παρόλο που θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες, όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος που μπορούμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Σιγητή, και για μία ακόμη φορά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σταβάρης, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Ε, όπως πάντα βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ αξιόλογη η έκθεσή του. Έχει κάνει αρκετές εκθέσεις και είναι όλες πάρα πολύ καλές. Έχει κάνει δύσκολη δουλειά ένα σημαντικό θέμα γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και αυτό μας το επιτρέπουν οι εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Είναι πάρα πολύ ισορροπημένη έκθεση και χαιρόμαστε μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε Κάποια κράτη-μέλη είναι σε διαφορετική κατάσταση, κάποια κράτη-μέλη έχουν 50% ανεργία των νέων, ενώ σε άλλες χώρες είναι 9%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως οι κοινωνικές επιπτώσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η πίεση προς τους νέους επίσης είναι διαφορετική. Η κατάσταση διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη, οι νέοι μεταναστεύουν λόγω του πολύ υψηλού επίπεδου ανεργία. Υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, Πορτογαλία και άλλες, όπου πάρα πολλοί νέοι φεύγουν από τη χώρα και δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί η κατάσταση παγιώνεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν σήμερα, δηλαδή αυτά του τομέα του ε, πολιτιστικού. Υπάρχουν τομείς όπως η δημοσιογραφία, η διαφήμιση, βιομηχανικό σχεδιασμός, αρχιτεκτονικοί τομείς που μπορούν να είναι το μέλλον, αλλά ε, ο κόσμος φεύγει μαζικά ε, στην περίπτωσή μας προς τη Βραζιλία και σε λίγα χρόνια είναι αυτοί δεν θα επιστρέψουν. Η οικονομία μας ως αποτέλεσμα αυτού θα γίνει λιγότερο βιώσιμη. Η οικονομία λοιπόν θα χωλαίνει. Όσοι έμειναν πίσω ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κάποια κατάρτιση, δεν έχουν πρόσβαση στην ε, αγορά εργασίας και θα αποτελέσουν βάρος μετά στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, άρα δεν θα είναι και τα οικονομικά βιώσιμα σε αυτά θα εστιάσω εγώ σε κάποιες από τις τροπολογίες που θα υποβάλω. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια πολιτική εστιασμένη σε περιφερειακό επίπεδο σε καιρούς κρίσης. Όλοι ξέρουμε τι έγινε μετά την ε, κρίση του χρέους στην Ευρώπη. Έχουμε ασύμετρα σοκ στην Ευρώπη και πρέπει να έχουμε άρα πολιτικές ως Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες θα καλύπτουν ναι ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με ε, ένα, μια γεωγραφική απόχρωση και διαφοροποίηση. Παραδείγματος χάρη. Να προσπαθήσουμε να δούμε το γεγονός το ότι κάποιες χώρες είχαν ε, μια κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και θα πρέπει ίσως να στηρίξουμε τοπικές αρχές και δήμους για να γίνουν π.χ. κάπου κόμβοι εταιριών βιομηχανικού σχεδιασμού ή αναλόγων ίσως και με κάποια στήριξη ενοικίου για να μπορέσουν οι εταιρείε να ανακάμψουν και να μειωθούν έτσι οι επιπτώσεις στους νέους κάτι το τελευταίο, όπως ε, και οι περισσότεροι συνάδελφοι, έτσι και εγώ μιλάω με πολλούς νέους ε, στην ε, χώρα μου και είναι αξιοσημείωτο το ότι παρά το ότι οι νέοι είναι αυτοί που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση, είναι οι περισσότερο φιλοευρωπαίοι. Αυτό με εντυπωσίασε πραγματικά. η μεγαλύτεροι ε, ωφελήθηκαν περισσότερο στα καλά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όμως έχουν έναν αισθηκτόδη αντιευρωπαϊσμό. Οι νέοι είναι διαφορετικοί, αντιλαμβάνονται πως η Ευρώπη είναι καλή για το δικό τους το μέλλον, αλλά θέλουν πραγματικά ένα εκδημοκρατισμό της Ευρώπης και θεωρώ πως με τις ιδέες που περιέχει έκθεση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε μια αμφίδρομη επικοινωνία από τους νέους προς την Ένωση και, και αντιστρόφως ουδέως. Γιατί νομίζω πως έχουν πολλά να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ταβάρης, κύριε euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τη συγκεκριμένη έκθεση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Δύο σημεία. Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε φυσικά πάντα τον στόχο αυτό της καταπολέμησης της εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα. Το πέρασμα από την κατάρτιση στην απασχόληση είναι θα έλεγα μια πολύ ευαίσθητη περίοδος και εκεί πάρα πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τις σπουδέ τους. Πρέπει λοιπόν να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και στην εκπαίδευση και στην απασχόληση και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Δεύτερον, έχουμε στόχους ποσοτικούς και ο κίνδυνος είναι να δημιουργήσουμε κάποια στάζ τα οποία είναι ε, μια μορφή απασχόλησης μόνο και μόνο για να κάνουμε στατιστικές θετικές. Όχι, τα στάζ που θα πρέπει να φτιάξουμε θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές προοπτικές. Να πω επίσης ότι σχετικά με τη στρατηγική για την νεότητα θεωρούμε ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλές εκθέσεις και πολλές προτάσεις για την νεότητα, έχουμε και τα προγράμματα ενημέρωσης, έχουμε τη στρατηγική για την νεότητα, έχουμε τις εγγυήσει για την νεότητα. Και σήμερα δύο υπουργοί απασχόλησης της Γερμανίας και της Γαλλίας συναντώνται και προτείνουν ένα νιου deal για την νεότητα στην Ευρώπη. Προ στιγμήν αυτό είναι γαλλογερμανικό, αλλά ο στόχος τους είναι να καλυφθεί το σύνολο της ζώνης ευρώ. Η ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, όπως και για το Εράσμους θα πρέπει να επιτρέψουμε στους νέους που σπουδάζουν να κάνουν στάζ σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτός της χώρας τους. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε όλα αυτά τα προγράμματα και δράσεις να λειτουργήσουν με συντονισμένο τρόπο γιατί αλλιώς θα, δεν θα αποφύγουμε επικαλύψεις και συγχύσεις. Λοιπόν, το νέο αυτό από τα δύο Υπουργεία είναι θετικό θα έλεγα γενικά. Θα πρέπει επίσης σαν βουλευτές να δούμε γιατί έχουμε τόσο λίγους νέους στο ημικύκλιο. Πράγματι ζούμε σε μια φάση πολιτική όπου όλα τα επίπεδα εξουσίας όπως και το κοινοβούλιο ε, θα έλεγα ελέγχονται από τους νέους αλλά δεν συνεργάζονται με τους νέους. Θα πρέπει να θέσουμε λοιπόν το εξής ερώτημα. Πώς ε, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις εμείς σαν βουλευτές σαν παράδειγμα στη Γαλλία και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα προς τους νέους. Θα πρέπει να αφήσουμε τις θέσεις για τους νέους και να μην μένουμε μετά τα 70 σαν παράδειγμα στο Κοινοβούλιο, να μην σορεύουμε τις πολιτικές εντολές, να ανοίξουμε εν περιπτώσει το δρόμο για τους νέους σαν πραγματικοί Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ πολύ. Αφήνεις τη θέση σου. Ευχαριστώ πολύ. Ας ε, εισαγωγούμε και κάποιες ποσοστώσεις ε, στις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αστείο είναι, αστείευομαι. Η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή. Ο συνάδελφός μας ειδικεύεται στις πολιτικές για τους νέους και πιστεύω ότι τώρα αυτή η εμπιστοσύνη που στην Ευρώπη γίνεται ορατή μέσω της πολιτικής για τους νέους. Έγιναν πολλά σφάλματα σε πολλές χώρες και τα συστήματα διαφέρουν. Παραδείγματο χάρη στη Γερμανία η ανεργία των νέων είναι στο 9%. Στην Ισπανία 50% πέρα από την ε, κρίση έγιναν και άλλα ασφάλματα σε διάφορα κράτη-μέλη. Λοιπόν, αυτή η στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική, πιο σημαντική τώρα μάλιστα. Πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση του συναδέλφου και πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρότατο μήνυμα προς τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των στατικικών. Σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχουν καν στατικικές. Και σε άλλα κράτη-μέλη έχουν ε, μπει στο χρονοτούλαπο και δεν έχουν εφαρμοστεί. Διότι αυτή η πολιτική των, ε, για τους νέους ε, διαιρείται με, ε, σε διάφορα υπουργεία. Πρέπει να στείλουμε μήνυμα λοιπόν στα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους. Υπάρχουν πολλές λύσεις που έχουν τονιστεί και αναφερθεί σε πολλούς τομείς. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Για το θέμα της χρηματοδότησης, όσον αφορά το έρασμος, την περιφερειακή πολιτική, τα διαθετικά ταμεία που χρηματοδοτούν την νεολαία, ε, υπάρχουν στρατηγικές, δεν υπάρχουν καλές στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν όμως σε επίπεδο 100 μελών. Και νομίζω ότι αυτή η έκθεση πρέπει να μας βοηθήσει να στείλουμε το ισχυρότατο μήνυμα προς τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν στρατηγικές, αλλά καμιά φορά αποτελούν μόνο δηλώσεις, δεν εφαρμόζονται, δεν υλοποιούνται. Θα πρέπει να απομιστούν τις ευθύνες στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε το Πρώτα απ' όλα επιτρέψατε μου να συγχαρώ τον κύριο Παπα-Νικολάου. Έχει προετοιμάσει ένα πάρα πολύ καλό κείμενο νομίζω πως έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς τη σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς είμαστε σε καιρό κρίσης. Ε, ξέρω πως οι νεότεροι άνθρωποι είναι και οι ασθενέστεροι. Διάβασα σήμερα πως ε, ε, προσφάτως πάνω από 300.000 Ισπανοί έφυγαν από την χώρα. Καταστροφικά δεδομένα. Όχι γιατί ε, δεν ε, πήγαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στη ΣΥΠΑ, στην Αυστραλία, σε άλλα μέρη του κόσμου. Πάρα πολλοί νέοι φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ζήτημα είναι αν θα επιστρέψουν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νέοι δεν, πάνε από... δεν φεύγουν μόνο από την Ισπανία. Ξέρουμε πως ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, δεν έχουμε αρκετούς νέους, πρέπει να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορούν να ζήσουν οι νέοι, οπότε τα κράτη-μέλη πρέπει βεβαίως να δουν το ζήτημα της μεταρρύθμισης αγοράς εργασίας. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κατάρτιση, η εκπαίδευση, έπρεπε να έχουν γίνει σοβαρότατε μεταρρυθμίσει του συστήματο εκπαίδευση πριν από πολύ καιρό. Έπρεπε να έχουμε επενδύσει ε, περισσότερο στην εκπαίδευση εδώ καιρό. Η Γερμανία είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώ μπορεί να μειωθεί η ανεργία των νέων μέσω ενό επιτυχού συστήματος εκπαίδευση. Ανησυχούμε ιδιαίτερα όλοι γιατί δεν έχουμε υπαρκεί οικονομικού πόρου για τον ε, τομέα τη εκπαίδευση. Αλλά σε καιρού κρίση πρέπει να αναρωτηθούμε το εξή χρηματοδοτούμε το εκπαιδευτικό σύστημα με τρόπο αποτελεσματικό, έχουμε δομήσει σωστά το σύστημα μας, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Υπάρχει χάσμα μεταξύ πανεπιστημίου και οικονομίας. Εάν έχουμε λοιπόν κάποια, κάποιο καλό σύστημα και μειωθεί αυτό το χάσμα θα μείνουν οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χειρότερο είναι πως η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει. Δεν τη βλέπουν οι νέοι όπως το παρελθόν. Οι νέοι δεν είναι πολύ ευρωσκεπτικιστές, αλλά αν δούμε διάφορες έρευνες βλέπουμε πως ο ευρωσκεπτικισμός υπάρχει στους νέους. Οι νέοι δεν έχουν ε, πολλές προοπτικές ε, αυτό φαίνεται να δείχνει και το τελευταίο ευρωβαρόμετρο. Οπότε πρέπει να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στους νέους. Αυτό θα γίνει βεβαίως αν αντιμετωπίσουμε τις αιτίες. Μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και του στήματος εκπαίδευσης. Ευχαριστώ κυρία Τομάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτήν την παρουσίασή του, την ιδιαίτερα ισόρροπη. Άκουσα από πολλούς συναδέλφους να λέγουν ότι θα πρέπει να στείλουμε προς τα κράτη-μέλη κάποια μηνύματα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε ο καθένας τα πράγματα του και τις υποθέσεις του και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής ε, πολύ σωστά αναφέρθηκε στις περικοπές ε, που έχουν προχωρήσει ορισμένες χώρες ε, στους προϋπολογισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και τις σοβαρές συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο για τους νέους. Πέραν τούτου όμως Αυτά τα, αυτές οι περικοπές συνδέονται άμεσα και με τις απαιτήσει της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης σχετικά με τους προϋπολογισμούς και την δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών. Δηλαδή ε, μείωση του χρέους και περικοπές που θίγουν τους προϋπολογισμούς, θίγουν θέματα όπως η ηλικία συνταξιοδότησης, ε, αυτό δεν το αναφέραμε, ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε τόσο πολλούς νέους ανέργους είναι ότι σε επίπεδο σταθερής ε, απασχόλησης το ότι αναγκάζουμε τους ε, μεγάλους ανθρώπους να εργάζονται όλο και περισσότερο σχετικά με τις ανάγκες του συνταξιοδοτικού, έτσι οι θέσεις ανοίγονται για τους νέους πολύ αργότερα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί, να βλέπουμε το σύνολο της εικόνας και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να κάνουμε μαθήματα στους άλλους όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε κάποιες αντιφάσεις στην δική μας πολιτική. Να προσθέσω εδώ ότι δυστυχώς δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία ορισμένων συναδέλφων γύρω από το φαινόμενο του ευρωσκεπτικισμού των νέων. Αυτό ίσχυε στη χώρα μου πριν κάποια χρόνια. Οι νέοι ήταν οι πιο Ευρωπαίοι και οι πιο δυναμικοί σε σχέση με την Ευρώπη. Σήμερα λόγω των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα πράγματα αλλάζουν. Και φοβάμαι ότι στις χώρες τις οποίες οι νέοι θα πρέπει να μεταναστεύσουν για να μπορέσουν να δουλέψουν, να δουλέψουν ο ευρωσκεπτικισμός θα γίνει βίαιος. Ε, σύντομα κύριε Ταβάρες. Ε, just very briefly, Σύντομα. Αντιλαμβάνομαι πως ε, από τη σκοπιά της Ένωσης βεβαίως γίνει διάκριση μεταξύ των νέων που φεύγουν από τη χώρα τους και μένουν εντός Ένωσης ή εκτός Ένωσης. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης εντός της Ένωσης, αλλά σε οικονομικούς όρους είναι το ίδιο. Δεν έχει διαφορά εάν ε, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί πάνε στη Βραζιλία ή στη Φιλανδία. Εάν οι χώρες του πυρήνα της Ένωσης δεν θέλουν να στηρίξουν την περιφέρεια για 10, 20, 30 χρόνια, πρέπει να φροντίσουμε τα, το φαινόμενο αυτό που είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ελεύθερη διακίνηση. Είναι ένα κενό, μια ολόκληρη γενιά φεύγει. δεν, πρέπει να υπάρξει. Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία που θα αποτρέψει, που θα επιτρέψει μάλλον σε αυτές τις οικονομίε οικονομίες να ισχυρές στο μέλλον ε, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ κύριο Σκαβαντό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος να πω ότι συμμερίζονται τα ουσιώδη των υποθέτων και αυτών που αναφέρω στην έκθεση και αυτά που υπογράμμισαν οι συνάδελφοι. Παρατήρηση έχω που δείχνει την μεγάλη σοβαρότητα του προβλήματος που ζούμε στην Ευρώπη και την αδυναμία των μέσων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων που είναι τραγωδία και έχει πάρα πολύ σημαντικές πολιτικές, ε, ε πολιτικές συνέπειες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι βλέπουμε τις προσπάθειες που γίνονται, κυρίως από κάποιες χώρες, αλλά τους λείπουν τα μέσα. Βλέπουμε άλλες προσπάθειες συνεργασίας που γίνονται, όπως της Γερμανίδας Καγκελαρίου με τον Γάλλο Πρόεδρο για το νέο deal όπως λένε διότι το νέο deal βασίζεται σε 6 δισεκατομμύρια δηλαδή 900, για εξαετία 900 εκατομμύρια ε, το χρόνο θα δαπανηθούν πιθανότατα στα 2-3 πρώτα χρόνια τα, τα χρήματα αυτά θα συζητηθεί και στον τρίλογο το θέμα αυτό το βράδυ Έχουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά χρειάζεται η στρατηγική για τους νέους τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χρημάτων και εγγύηση δανειοδότηση από τις διεθνείς αγορές. Τα δημοσιονομικά των χωρών του Νότου είναι που ε, έχουν πρόβλημα και δεν μπορεί ο τομέα να έδωσε την εγγύηση. Είναι νομικό πρόσωπο η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να κινηθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τα μέσα που διαθέτει. Δεν έχουμε δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα ε, της ανεργίας των ε, νέων. Ε, λοιπόν, απελπίζονται οι νέοι και δημιουργούν ε, μια, μια πολιτική διαφορία εξ αυτού. Σαντιάγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως η δική μου χώρα να είναι η χώρα της Ευρώπης όπου το πρόβλημα της ανεργίας των νέων είναι μάλλον το σοβαρότερο. Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία. Πολλά λέγονται γύρω από αυτό, πολλά λέγονται για πιθανές λύσεις, μιλάμε για τον ρόλο φυσικά της εκπαίδευσης που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πρέπει να επιμείνουμε στα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει ζωτική σημασία και θα πρέπει επίσης να δώσουμε περισσότερη αξιοπρέπεια και βάρος στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πολλοί νέοι ε, μετά τις σπουδές τους συνεχίζουν να σπουδάζουν διότι γνωρίζουν ότι δεν έχουν δυνατότητα απασχόλησης. Η μοναδική λύση δυστυχώς είναι η οικονομική ανάκαμψη. Όχι δυστυχώς είναι η δυνατότητα η οικονομική ανάκαμψη. Αλλιώς οι νέοι και οι νέες θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε τις πολιτικές της ανάκαμψης της οικονομίας, η λιτότητα έχει κάποια όρια και γίνονται πολλές συζητήσεις γύρω από αυτό, αλλά μια απόλυτη επιδίωξη της οικονομικής λιτότητας δεν οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχει πάρα πολύ σημασία λοιπόν να αναζητήσουμε πολιτικές που θα βοηθήσουν να, να ανακάμψει η πολιτική να ασκήσουμε και πολιτικές, να εφαρμόσουμε συγγνώμη και πολιτικές λιτότητας όπου είναι απαραίτητο, αλλά να αναζητήσουμε κάποιες νέες λύσεις, γιατί αυτές μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Η μοναδική λύση είναι οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προκόψουν και να δώσουν θέσεις εργασίας στους νέους. Ο κύριος Λεζόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, είπε και ο εισηγητής σας, η έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής έχει σαν στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής για την νεότητα για τον πρώτο κύκλο μέχρι το 18 και να προτείνει προτεραιότητες δράσης ε, για τα τρία αυτά χρόνια, το δεύτερο κύκλο δηλαδή 15-18 ασυνοδεύεται άλλωστε από δύο έγγραφα τα οποία δίνουν πολλές πληροφορίες για την κατάσταση των νέων σε διάφορες χώρες και για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από διαφορετικές χώρες και τους άξονες της στρατηγικής ε, για την νεότητα τα πρώτα χρόνια. η βασική στόχοι αυτής της στρατηγικής για την νεότητα είναι δύο. Καταρχάς θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και στην απασχόληση και στην εκπαίδευση και πολλές παρουσιάσεις σήμερα ε, επέμειναν σε αυτό. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε τη συμμετοχή των νέων στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στην κοινωνία. Η πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε ορισμένες χώρες συνδέεται με την πολύ σημαντική ανεργία και η έκθεση περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ορισμένες χώρες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι' αυτό. Η σημασία, το βάρος αυτής της άσχημης κατάστασης δείχνει και εξηγεί ότι και για τη δεύτερη τριετή περίοδο έχουμε υπογραμμίσει και μένουμε στις συνέπειες της ανεργίας για τους νέους και όχι μόνο στην πρόσβαση στην απασχόληση. Τίθεται λοιπόν το θέμα του μη αποκλεισμού των νέων, της υγείας και της ευημερία των νέων. Στην παρούσα περίοδο επιμένουμε σε θέματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων που ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται, τα λεγόμενα νίτς. Εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα τους το ταχύτερο δυνατόν και κατά προτεραιότητα. Όπως έλεγα η στρατηγική στην οποία αναφερόμεθα είναι σφαιρικού τύπου. Δεν περιορίζεται σε θέματα απασχόλησης και εκπαίδευσης αλλά και σε άλλους τομείς όπου έχει υπάρξει πρόοδος. Σαν παράδειγμα στην συμμετοχή των νέων ή στα θέματα της εθελοντικής απασχόλησης που έχει τεθεί το θέμα σήμερα το πρωί. Η έκθεση αναφέρεται σε κάποιες ε, αντιλήψεις που υπάρχουν σχετικά με την εφαρμογή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη στρατηγική. Αναφέρθηκε σαν παράδειγμα το επόμενο πρόγραμμα στον τομέα της κατάρτισης της νεότητας και του αθλητισμού που περιλαμβάνει δράσεις και σχετικά με τις μη τυπικές παραδοσιακές μορφές ε, ε, εκπαίδευσης Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης και αυτό αναφέρθηκε επίσης το πρωί την σημασία της διατομεακής διυπουργικής συνεργασίας είναι προϋπόθεση σε πολλές χώρες για την διασφάλιση των πολιτικών για την νεότητα. Υπογραμμίζεται επίσης η σημασία να υπάρξουν ποιοτικά στάζ, τα οποία να μην είναι στάζ αυστηρά προσωρινής απασχόλησης. Ο εισηγητής σας σωστά υπογραμμίζει την σημασία που θα πρέπει να δώσουμε σε ορισμένα τα μέσα, από τα μέσα που περιλαμβάνονται στη στρατηγική. Ο διαφρομένος διάλογος, σαν παράδειγμα. Να σημειώσουμε ότι αυτή την εβδομάδα υποδεχόμαστε εκπροσώπους των νέων από όλε τις ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να υπάρξει μια επανεξέταση του διαφρωμένου διαλόγου όπως τέθηκε σε εφαρμογή τα προηγούμενα τρία χρόνια, για να καταστεί πιο αποτελεσματικός και να λάβουμε υπόψη μας και τις γνώμες των νέων. Υποστηρίζουμε αυτά που υπόθηκαν σήμερα το πρωί και για τον ρόλο των οργανώσεων που εκπροσωπούν τους νέους και σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, αλλά και σχετικά με την ανάπτυξη των προσωπικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων των νέων γιατί πολλές φορές σε επίπεδο οργανώσεων νέων ε, αναπτύσσονται ε, και τα θέματα που έχουν σχέση με την μη τυπική, μη επίσημη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τέθηκε επίσης ε, και το θέμα της συμμετοχής των νέων στα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Εμείς δημοσιεύσαμε μία μελέτη την προηγούμενη Παρασκευή στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τους Νέους που δεν έχει τελειώσει ακόμα θα δείτε πληροφορίες ενδιαφέρουσες, αντιφατικές μερικές φορές αναχώρα, αλλά που δείχνουν ότι στους νέους εξακολουθούν να πιστεύουν στην Ευρώπη περισσότερο από ό,τι σε άλλες κατηγορίες ηλικιακές. Ε, στην έκθεση του κυρίου Παπα-Νικολάου υπογραμμίζουμε και την σημασία που έχει να βελτιώσουμε ε, τις γνώσεις που έχουμε για την πραγματική κατάσταση των νέων, για την ανάγκη χρήσης καλύτερων στατιστικών, για μια καλύτερη γνώση των νέων γενικότερα, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και εργαζόμαστε γι' αυτό με τη Eurostat. Ο εισηγητής σας ε, υπογραμμίζει επίσης και ένα θέμα το οποίο δεν είναι άμεσα ένα μια γραμμή δράσης της στρατηγικής για την νεότητα, αλλά που έχει σημασία και το συναντάμε σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής της στρατηγικής, τις νέες τεχνολογίες και τα νέα μέσα. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γύρω από θέματα όπως η προστασία των νέων και σας σημειώνω εδώ ότι δημοσιεύσαμε μια μελέτη πρόσφατα για νέους τρόπους συμμετοχής των νέων στην Ευρώπη που υπογραμμίζουμε ακριβώς τις δυνατότητες τις οποίες ε, ανοίγουν τα νέα μέσα για τη συμμετοχή των νέων. Πάντα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και κυρίως σε σχέση με το τι μπορεί να προσφέρουν στον τομέα της εκπαίδευσης να πω ότι ε, η Επίτροπος Βασιλείου και άλλος ένας Επίτροπος θα ξεκινήσουν ε, τον επόμενο μήνα μια νέα πρωτοβουλία για τη σωστή εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Ε, το πρόγραμμα αυτό θα ονομάζεται Opening Up Education. Λοιπόν, και σε αυτό το θέμα και σε άλλα είμαστε στη διάθεση του εισηγητή σας αν τυχόν χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ κύριε Λεζόν. Ήθελα πω ακόμη μια φορά. Κύριε Φίσα, βεβαίως χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας, αλλά αυτό σημαίνει και ε, εκπαιδευμένους νέους. Είναι φαύλος κύκλος δηλαδή. Το πρόβλημα είναι πως σε πολλές χώρες εδώ και χρόνια το θέμα της σωστής επαγγελματικής κατάρτιση δεν αντιμετωπίστηκε. Δηλαδή, έλεγαμε στους νέους πως ε, θα κάνετε κάτι μόνο αν πάρετε ακαδημαϊκό απολυτήριο και σπουδάσετε. Και μετά μας λείπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι για τις επιχειρήσεις και μετά δεν υπάρχουν επιχειρήσεις γιατί λείπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Δηλαδή, Είμαι εδώ πέρα 25 χρόνια. Στη δεκαετία του 90 προσπαθούσα πάντα στις συζητήσεις να πω πως το θέμα της ανεργίας των νέων συνδέεται στενά με ε, ένα λανθασμένο προσανατολισμό των νέων ε, όσον αφορά την πολιτική της εκπαίδευσης. Γιατί στη Γερμανία έχουμε τόσο χαμηλή ανεργία των νέων. Βεβαίως, εντάξει, είναι και καλύτερα τα πράγματα από πλευράς θέσεων εργασίας, αλλά δεν είναι αυτό το μόνο. Αν είχαμε τόσους πολλούς νέους με, όπως οι Ισπανοί που έχουν βγάλει το πανεπιστήμιο αλλά δεν έχουν ε, πρακτική εκπαίδευση, θα είχαμε και εμείς πολύ ψηλότερη ενέργεια των νέων. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε νέους τρόπους στο θέμα της ε, κατάρτισης. Και αυτό το κάνουν και οι Ολλανδοί και οι Αυστριακοί και άλλοι. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αυτή την διπλή οδό. Κατάρτιση και στην επιχείρηση και στο σχολείο ταυτόχρονα. Και στο τέλος έχει κάποιος πραγματική δουλειά στα χέρια του με την οποία μπορεί κάτι να κάνει. Και άμα θέλει αργότερα να σπουδάσει και παραπέρα. Η ιδέα αυτή είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η Ισπανική κυβέρνηση θέλει και ενδιαφέρεται να συζητήσει το θέμα αυτό με την Γερμανίδα Υπουργό Απασχόλησης. Συνεργάζονται, νομίζω. Ε, δεν θα οδηγήσει βεβαίως αυτό αύριο στην Ισπανία σε χαμηλότερη ανεργία των νέων, αλλά σε βάθος χρόνου. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι μια πολιτική που δεν πρέπει να προσανατολίζεται στις εκλογές αλλά να προσανατολίζεται στο μέλλον. Οπότε υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Θα ήθελα επίσης να πω πως έχουμε πολύ μικρότερους τομείς και Κοιτάξτε, να σας πω και για τους Γάλλους ε, συναδέλφους. Εγώ μένω στο Ζάρλαντ ε, και ποιο είναι το πρόβλημα. Εμείς είμαστε στα σύνορα με Γαλλία και Λουξεμβούργο και δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν νέους. Ο κομμωτής με κουρεύει, δεν μπορεί να πάρει Γάλλους νέους να τους μάθει τη δουλειά γιατί πρέπει να πληρώνει κάποιο ειδικό φόρο στο γαλλικό κράτος. Τρελή κατάσταση. Σκεφτόμαστε τώρα με διαφόρους ε, ειδικούς πώς θα λύσουμε αυτό το διμερές ε, πρόβλημα. Και μου στέλνουν email και μου λένε «Μα δεν είναι Ευρώπη αυτή, ο γιος μου δεν μπορεί να πάει στο Ζάρλαντ να κάνει την πρακτική του άσκηση» και μιλάει γερμανικά. Γιατί η γιαγιά μιλούσε μια γερμανική διάλεκτο. Ε, είναι Ευρώπη αυτό. Όχι. Πρόκειται για ένα διμερές πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε. Και πρέπει να το λύσουμε προς το συμφέρον της νέας γενιάς. Ναι, αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς εδώ αυτά τα προβλήματα, αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω, το κείμενο του συναδέλφου του κυρίου Παπα-Νικολάου είναι μια ανασκόψη του τι έπρεπε να έχει γίνει από το 2010 μέχρι το 2012. Για το μέλλον πρέπει βεβαίως να φροντίσουμε και να δούμε πως ε, και η Κομισιόν έχει κάνει κάποια πράγματα. Και το Συμβούλιο έχει αυτή την πρωτοβουλία, πώς λέγεται, ε, πρωτοβουλία για την εκπαίδευση της νεολαίας, όπου δίνει 3 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια ευρώ για το θέμα αυτό. από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κάτι το οποίο δείχνει πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να γίνουν αυτές οι συνδέσεις. Ε, λέτε πως δεν θα μας ε, σώσουν αυτά. Ε, μα δεν θα μας σώσει τίποτα, αλλά λίγα λίγα πραγματάκια από εδώ και από εκεί και μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε νομίζω μια καλύτερη κατεύθυνση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αλλιώς θα πάει πραγματικά μια γενιά χαμένη. Και μετά αναφέρομαι σε αυτό το οποίο είπατε το θέμα δηλαδή του εάν οι νέοι είναι σε θέση να ανοίξουν μόνο τους μία επιχείρηση, αν είναι αρκετά δημιουργική. Το συζητήσαμε και με την έκθεση της Μαρή Τερέζ. Λείπει κάπου το, το θάρρος, αν θέλετε, να, να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση. Ίσως ήταν πολύ απλό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έβρισκε κάποιος μια θέση εργασίας, ε, το κρατούσαν ε, στη ζωή επιδοτήσεις. Εάν αναγκάζονταν να κάνει κάτι, κάτι το οποίο συμβαίνει στην Αμερική γιατί δεν έχουν κάποιο κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας, υπάρχει και περισσότερη δημιουργικότητα. Γι' αυτό θα ήθελα να δούμε το θέμα της δημιουργικότητας περισσότερο στην ε, νεολαία. Γιατί έτσι νομίζω οι νέοι θα μπορέσουν να, να βρουν ή να δημιουργήσουν μια δουλειά. Αυτά από μένα. Θα ήθελα να ξαναδώσω τον λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου. Ε, και κάτι ακόμα. Μέχρι την Πέμπτη πρέπει να έχουμε υποβάλει τις τροπολογίες. Ε, λυπούμε, αλλά μας ε, έκανε η Επιτροπή Απασχόληση να περιμένουμε. Γεώργια. I believe today's Πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι όλοι μας ενδιαφερόμαστε πολύ για την κατάσταση των νέων και βέβαια πιστεύω ότι ένα ακόμα συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βοηθήσουμε τους νέους όλων των κρατών μελών. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με την παρούσα κατάσταση. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που περνά μια περίοδο ύφεση. Έχουμε όλες αυτές τις περικοπές των προϋπολογισμών και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Έχουμε αυτή την απογοήτευση των πολιτών μας και αυτό συνδέεται και με τον ευρωσκεπτικισμό όπως αποκαλείται και που αναφέρθηκε όλα αυτά τα συναισθήματα δεν είναι πολύ αισιόδοξα. για τις ε, προοπτικές, για τις ευρωπαϊκές ιδέες μας και τις ευρωπαϊκές αξίες. Προβληματιζόμαστε για το πώς θα μπορούμε να, μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή την έκθεση. Θα θυμόσαστε ότι στην αρχική μας εισαγωγή, εδώ και μερικούς μήνες, επικρίναμε τα αποτελέσματα των κατών μελών, την αποτελεσματικότητα των στατηγικών. Αλλά πρέπει σήμερα να παραδεχτούμε ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια στατηγική και αυτό άλλωστε συζητήσαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι γεγονός ότι υπάρχει στρατηγική. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια στρατηγική και είναι εξίσου πολύ σημαντικό ότι σήμερα συζητούμε την πρόοδο στρατηγικής. Βλέπουμε και αποτιμούμε το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πώς μπορούμε να ε, συμβάλλουμε μέσω ιδεών και προτάσεων στην αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ακούμε πολλά. Επαναλαμβάνω ότι σε... ακολουθούμε πρωτοβουλία σε επίπεδο Συμβουλίου και θα αναλυφθεί η πρωτοβουλία τον επόμενο μήνα και προβλέπεται η συγκεκριμένη συνεδρίαση για το θέμα. Και ο πρόεδρος Μπαρόζο πριν από δύο χρόνια περίπου είπε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για την νεολαία. Βλέπουμε τις ομάδες κρούσης των κρατών μελών. Δεν τροφοδετούμε θα μα πληροφορήσουν αυτά τα επιτεύγματά τους σε οποιοδήποτε τομέα δράσεως χρειάζεται διατομεακή προσέγγιση, οριζόντια. Διαφορετικά τα θέματα των νέων δεν μπορούν να λυθούν αποτελεσματικά. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμόσαστε εσείς, Κυρία Πρόεδρε, πριν από μερικούς μήνες έγινε μια συνάντηση, διοργανώσαμε μια εκδήλωση με τη συμμετοχή δική σας και του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας. Ξανασυζητήσαμε το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα προγράμματα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους και κυρίως στις χώρες που είναι στο επίκεντρο της κρίσης. Ισπανία, Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Και εισήγαγα το θέμα, είπα ότι έχουμε 50-60% ανεργία των νέων, η Γερμανία έχει 8, 9, 10% ανεργία των νέων και τότε έρθει η σειρά σας και είπατε ναι, αλλά στη Γερμανία έχουμε διτό σύστημα και ήταν πολύ εύκολο να το πείτε αυτό. Και πρέπει να σας πω όμως την επόμενη μέρα, κα... την επόμενη μέρα στα ελληνικά μέσα δύο-τρεις δημοσιογράφοι έγραψαν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν χρησιμοποιήσουμε το σύστημα, διότι πιθανότατα μπορούμε να έχουμε εργο, εργαζομένους χωρίς να έχουν προστατευμένα δικαιώματα στον αφορά απασχόληση. Δεν είναι αλήθεια, είναι προκατάληψη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στους λαούς μας. Θα πρέπει να εστιαστούμε επί των λύσεων και να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι αν δεν αλλάξουμε μυαλά αν δεν προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών, εάν δεν δούμε το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα μέσα, τότε θα παραμείνουμε σε συζήτηση θεωρητικού επίπεδου χωρίς προστιθέμενη αξία. Πιστεύω ότι όλα τα ζητήματα που αναφέρονται είναι αρκετά σημαντικά, όπως η διαρροή εγκεφάλων και η συζήτηση που αφορά τη χαμένη γενιά, την παρούσα γενιά που δεν μπορεί να είναι χαμένη, θα μπορούσε μάλλον να είναι χαμένη γενιά αν δεν προσέξουμε ε, όσον αφορά τις πολιτικές μας. Κανείς δεν μπορεί να είναι αισιόδοξο και σίγουρος ότι σύντομα θα έχουμε αποτελεσματικές λύσεις και αποτελέσματα που θα επιφέρουν τη μεγάλη αλλαγή σε σχέση με αυτά που γίνονται σήμερα. Αν δούμε τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, ε, όλοι θα συμφωνούσαμε. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι όσον αφορά την ουσία των θεμάτων είναι να είμαστε όσο πιο καινοτόμοι μπορούμε, όσο πιο δυναμικοί μπορούμε. Γι' αυτό αναφερθήκαμε στις νέες τεχνολογίες και στα κοινωνικά μέσα στην έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πού βρίσκονται οι νέοι αυτή την περίοδο. Πώς μπορούμε να τους πλησιάσουμε. Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι παρόλο που έχουμε πολύ σύντομη περίοδο υποβολή τροπολογιών. Οι συζητήσεις θα είναι πολύ καρποφόρες και ο συντονισμός. Στις τελευταίες διαπραγματεύσεις επί των τροπολογιών πιστεύω ότι όλες οι τροπολογίες μπορούν να θεωρηθούν πρόσδεκτες. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι αποτελεσματικό. Καινοτόμο. Ιδέες, λύσεις για τα προβλήματα των νέων. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για μία ακόμη φορά, για τα καλά τους σχόλια, για την συνεισφορά τους. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπόρις που είπε ότι θεωρούμε σαν κάποιος που γνωρίζει το πώς αντιμετωπίζω τα θέματα της νεολαίας. Ήθελα να του πω ότι έχω γκρίζα μαλλιά αυτές τις μέρες. Και τα γκρίζα μαλλιά είναι περισσότερα από πολλών συναδέλφων. Προσπαθώ να παρακολουθώ τις εξελίξεις, προσπαθώ να είμαι όσο πιο αποτελεσματικός γίνεται, ελπίζω αυτό να σας αρκεί, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην τελική ψηφοφορία της εκθέσεως. Είναι καλός ο χρονισμός για την έκθεση, καθοδόν προς το Συμβούλιο και πιστεύω θα αποτελέσει μια πολύτιμη συνεισφορά, καλό μήνυμα που θα προέρχεται από, τη, από το Ευρωκοινοβούλιο προς όλους τους θεσμούς των κρατών μελών για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Όσο γνωρίζετε όλοι, η 5η στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Καλώς. Ερχόμαστε στο σημείο 6, αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ενδεχόμενες διέξοδοι. Συνέχιση δηλαδή της τελευταίας συζητήσεως, διότι συνεχίσαμε, συνεχ, συζητούν περισσότερο την ανεργία από ό,τι άλλο είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Ντελβάλη προς την, όσον αφορά το έγγραφο της Επιτροπής Απασχόλησης. Θα είναι συντομότερη η συζήτηση. Καλύψαμε το θέμα. Παρουσιάστε όμως την γνωμοδότηση. Ο κύριος Ντελβάλη λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πράγματι έχετε δίκιο. Αυτή η γνωμοδότηση που παρουσιάζω ε, συνδέεται λογικά με την έκθεση του κυρίου Παπα-Νικολά, αυτό είναι σίγουρο. Άλλη παρατηρήση, πριν μπω στην ουσία, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τις σκέψεις που εκφράσετε εσείς στην αρχή, κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά το θέμα και κυρίως με αυτό που μπορούμε να αποκαλέσουμε τη θεωρία του φαύλου κύκλου, διότι σίγουρα αυτός ο φαύλος κύκλος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ε, για την επίλυση αυτής της τραγωδίας που εξετάζουμε. Να μπω τώρα στην ουσία, α, κατά τη δική μου άποψη και α, κατά την άποψη του τομέα της παιδείας, κάνω τέσσερις συστάσεις που πιστεύω ότι μπορούν να καταπολεμήσουν το δράμα αυτό της ανεργίας των νέων που όλοι αντιμετωπίζουμε και πλήττει το 23% του πληθυσμού των νέων της Ευρώπης και σε κάποιες χώρες όπως η Ισπανία ή η Ελλάδα μπορεί να φτάσει πάνω από το 50% ενεργεία των νέων. Προτείνω μια αύξηση ε, ε, της χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης των κρατών μελών και διτό ποιοτικό ε, σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης. Ποιοτικό, είναι σημαντικό αυτό που γραμμίζεται. Χρειάζεται επικύρωση της μόρφωσης ακαδημαϊκής και μη και πρέπει να ενισχύσουμε την πρωτοβουλία για την εγγύηση για τους νέους. Όσον αφορά την πρώτη σύσταση, θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου όσον αφορά τις περικοπές του προπολογισμού που πραγματοποιούνται σε επίπεδο κρατών μελών στον τομέα της παιδείας. Ε, θα, θα, πρέπει, θα πρέπει να, παίξει ρόλο σημαντικό η εκπαίδευση όσον αφορά την ενεργεία των νέων και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι από πλευράς προπολογισμού για την παιδεία. Ε, θα πρέπει να υπάρξει παιδεία για να αυξηθεί και η ευμάρεια η κοινωνική. Ε, δεν υπάρχει λύση ποιοτική αν δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Λοιπόν, επένδυση όσον αφορά την κατάρτιση, στην εκπαίδευση, σε, το, σε αυτή την περίοδο της κρίσεως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί από της εθνικής κυβέρνησης σαν κόστος, αλλά περισσότερο σαν μια επένδυση, αναγκαία επένδυση ε, και ανεκτήμητης αξίας που θα επιτρέπει στους νέους να έχουν ένα μέλλον. Μετά θα πρέπει να χτυπήσουμε τον κόδωνα του κινδύνου προς τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα διτό σύστημα κατάρτισης. Όλοι το ζητήσαμε, να δούμε αν θα καταφέρουμε ε, να το πετύχουμε, ε, να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημά μας. Λοιπόν, συνδυάζοντας την, τη τα θεωρητικά μαθήματα και τα πρακτικά, αν γεφυρώσουμε την κατάρτιση και την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε να αποκτώνται άμεσες δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας μέσω διαφόρων επαγγελματικών προσόντων ε, παρά όμως τα θετικά αποτελέσματα της διπλής επαγγελματικής κατάρτισης όσον αφορά το, τη μείωση της ανεργίας πιστεύω ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει να σέβεται κάποιο κώδικα συμπεριφοράς ε, ποιοτικό για να ε, δημιουργούνται συνθήκες για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τους νέους, να καταργηθεί ε, η ε, επισφαλής εργασία που υπάρχει τώρα στην αγορά Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια χέγγια που θα θεσπιστούν. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας. Και εγώ υποστηρίζω την επαγγελματική κατάρτιση. Μετά όσον αφορά αυτά που είπατε κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είμαι υπέρ της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο κ. Ζόχαν Μπούντενμπροκ που ανέφερε ο Τόμας Μαν στο βιβλίο του η Μπούντενμπροκ η, ε, μια οικογένεια η παρακμή μιας οικογένειας ε, δείχνει πολύ καλά το θέμα αυτό ε, εγώ έχω αντίθετη άποψη όμως όσον αφορά το σύμβουλο Μπούντεμπρουκ. Λέει λοιπόν εκεί ο Μπούντεμπρουκ στο βιβλίο ότι, ότι ιδεά, αναφέρει κάποιες ιδεώδεις πρακτικές με τις οποίες όμως εγώ δεν είμαι σύμφωνος. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τη σωστή κατάρτιση. Τα πτυχία τα κλασικά θεωρούνται ε, σαν περιτά. Είναι σαφές λοιπόν ότι από την πλευρά μας ε, είναι ανόητη προσέγγιση που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα. Ο σύμβουλος λοιπόν ήταν αντίθετος όσον αφορά τα ωφέλη της διπλής επαγγελματικής κατάρτισης. Ε, προτιμούσε την εγκατάλειψη της κλασικής εκπαίδευσης. Πιστεύω ότι είναι συμβατά και τα δύο. Η επένδυση στην επαγγελματική κατάρτιση δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος της ανώτερης εκπαίδευσης και εδώ απαντώ στο σύμβουλο σε αυτά που λέει στο εν λόγω βιβλίο είναι ένα μέσο θεμελιώδου σημασίας για να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια οικονομία της γνώσης που θα είναι ανταγωνιστική και η οποία θα δρά με δυναμικό τρόπο και θα κινείται στον κόσμο όπως αναφέρεται και στατηγική του 2020. Τρίτον, συστήνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την αναγνώριση των προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και πιο συγκεκριμένα μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, των βαθμολόγησης πιστώσεων που δίνονται αν θέλετε, αναγνώριση όσον αφορά τα προσόντα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα ε, αναγνώρισης των τίτλων στην ανώτερη εκπαίδευση και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την κατάρτιση, τη μη πανεπιστημιακή. Αυτός που έχει σημαντικές γνώσεις θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται για να έχουμε δυναμική οικονομία. Η εγγύηση για τους νέους. Απευθύνω έκκληση προς τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη να αυξήσουν το ποσό των 6 δις ευρώ προβλέπεται για το 2014-2020 και εφαρμογή της ε, πρωτοβουλίας ε, ε, εγγύηση για τους νέους που θα φτάσει μέχρι 30 χρόνια. Όσον αφορά τις τροπολογίες θα μπορούσα να λάβω και άλλες, ε, υπόψη μου άλλες ιδέες που δεν είχα χρόνο να παραθέσω. Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω διάφορα στοιχεία συγκεκριμένα πρακτικής φύσης που μπορούν να είναι ενδιαφέροντα για σας. Καταρχάς πρέπει να προσέξουμε διότι η ομάδα προβληματισμού σήμερα στο Παρίσι εξετάζει, συζητά το θέμα της ανεργίας των νέων. Σήμερα η κυβέρνηση, η γαλλική κυβέρνηση στο Παρίσι θα υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά την ενεργεία των νέων και έχω και ένα άλλο σχόλιο. Πόσους πόρους, τι χρήματα διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο αυτό, την ενεργεία των νέων. Ας κάνουμε υπολογισμούς, επί χάρτου, θεωρητικά, διαθέτουμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στα αποθεματικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014-2020. 16 εκατομμύρια επιχάρτου πόρους που δεν χρησιμοποιήθηκαν ακόμα. Και θα ρισκάρω να πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα 10 δισεκατομμύρια που η Δημόσια Γερμανική Τράπεζα η Δημόσια Τράπεζα με το FW, ε, FW, τα αρχικά θα μπορούσε να διαθέσει για επενδύσεις για το μέλλον. Θα μπορούσε, λέγω, για το μέλλον της Ευρώπης. Συνολικά, επί χάρτου, 32 δισεκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση του σοβαρότερου προβλήματος της Ευρώπης. Μέχρι τώρα όμω δεν υπάρχει κανένα προγραμματισμό και από πλευρά των κρατών μελών και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τίποτα δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Και η Γερμανία, τη οποία την βούληση την χαιρετίζω, δεν έχει δώσει κάτι συγκεκριμένο. Μια και η Γερμανία ήταν πρωταγωνίστρια σε αυτά τα οποία έλεγε η Πρόεδρος προηγουμένως, τι πρωτοβουλίε που αναλαμβάνει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, δηλαδή για τη συνεργασία με άλλες χώρες μέλη, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που προχωρήσει με αυτά τα οποία λέγει, αυτό θα συναντήσει κάποια εμπόδια θα έλεγα διακανονιστικά τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. θα πρέπει καταρχάς να περάσει από την αρμόδια επιτροπή της Ομοσπονδιακής Βουλής. Στις 3 Ιουλίου στο Βερολίνο έχει συγκληθεί μια συνάντηση στην οποία είναι προσκεκλημένοι η Υπουργή Γεωργίας ε, των 27 χωρών και των ε, αρμόδιων Υπουργείων των 27 χωρών, έτσι ώστε να συμφωνηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο στις 3 Ιουλίου στο Βερολίνο με συγκεκριμένες μορφές χρηματοδότησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως ανοίγει ένα επιπλέον πρόβλημα. Η Ομοσπονδιακή Βουλή δεν θα μπορέσει να το εκρίνει σε αυτή την τελική φάση της ε, ε, νομοθετικής περίοδου, γιατί η τελευταία συνεδρίαση πριν από τις διακοπές θα είναι 27 Ιουλίου. Ιουνίου, συγγνώμη, πριν από τη συνάντηση της 3 Ιουλίου. Το Σεπτέμβριο προβλέπονται συναντήσεις στις 2 και στις 3 Σεπτεμβρίου που φυσικά θα ασχοληθούν με, με θέματα υποεκκρεμότητα και μετά θα ακολουθήσουν οι προετοιμασίες για τις ομοσπονδιακές εκλογές. Συνεπώς λοιπόν ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει τίποτα συγκεκριμένο και μέχρι το φθινόπωρο δεν προβλέπεται να υπάρξει κάτι το συγκεκριμένο. Εγώ θα καταλήξω σε κάτι το οποίο ακούγεται σκληρό αλλά δεν το λέω εγώ. Η Bill Zeitung το 2008 χαρακτήρισε την τράπεζα αυτή ε, την πιο ανόητη τράπεζα της χώρας γιατί είχε μεταφέρει 350 εκατομμύρια ευρώ στη Lehman Brothers. Λίγες ώρες πριν η Lehman Brothers ε, αναφλεγεί και καταλήξει σε πτώχευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν μας δείχνει σε τι φαύλο κύκλο βρισκόμαστε κυρία Πακ. Δείχνει όμως και τι προκάλεσε την κρίση αυτή στην οποία παλεύουμε τώρα και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε τους νέους με αυτές τις πρακτικές. Να σχολιάσω μια φράση στην οποία αναφερθήκατε σχετικά επίσης και τους Μπούντεμπροκ, το βιβλίο του Τόμας Μάν. Αγαπητέ κύριε Δελβάλε, εγώ δεν εκπροσωπώ την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αλλά δεν συμφωνώ απολύτως και για το ότι φταίει η Γερμανία για το εκπαιδευτικό σύστημα της ε, Ισπανίας. Αν είναι να βοηθήσουμε, το κάνουμε και προς το δικό μας συμφέρον, γιατί θέλουμε πραγματικά οι Ισπανοί να βρίσκουν δουλειές στην Ισπανία. Και είμαι σίγουρη, καμία γερμανική βουλή ανεξαρτήτως σύνθεσης δεν θα είχε καμία αντίρρηση. Ε, η Υπουργό ε, Εργασία ε, μαζί με τη δική σα Υπουργό να, συνεργαστούν. Ανεξαρτήτω του ποιο κυβερνάει, είτε κυβερνά το δικό μου κόμμα, οι χριστιανοδημοκράτε ή οι δικοί σα οι φίλοι, οι σοσιαλδημοκράτε. Ε, είστε σίγουροι ότι οι Γερμανοί βουλευτές είναι λογικοί και χαίρονται τα λεφτά να μην πηγαίνουν στις τράπεζες αλλά σε πρωτοβουλίες που προωθούν την εκπαιδευτική κατάρτιση των νέων. Οπότε σε αυτό συμφωνούμε. Και είμαι σίγουρη, γνωρίζω την, ε, την κυρία Υπουργό. Νομίζω θα τα καταφέρει. Είτε είναι η διαδοχό της ε, κάποια σοσιαλδημοκράτης, είτε όχι, θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Αυτά περί Γερμανίας ε, και Ισπανίας και του χρέους και της, ευθύνη ευθύνης των Γερμανών για την κρίση. Λοιπόν, κυρία Σαντζεσμιτ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Μενέντε Δεβάγια για μια συγκεκριμένη έκθεση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη εδώ. Έχει τεθεί το θέμα για τι πιστώσεις έχουμε στη διάθεσή μας. Να πω ότι υπάρχουν τα διαφορετικά ταμεία. Να θυμίσω ότι η στρατηγική για την νεότητα, όπως ε, δείχνει και η έκθεση του κυρίου θα αναπτυχθεί και σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Το κοινωνικό ταμείο θα παίξει ένα ρόλο, θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση των νέων, για την επιστροφή στην απασχόληση ή για την πρώτη απασχόληση. Και να θυμίσω επίσης ότι οι στρατηγικές αυτές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές που έχουν τους μοχλούς δράσης. Σε ορισμένες χώρες είναι υπεύθυνε και συνεργάζονται με τον επιχειρηματικό κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε όπως μπορούμε τις στρατηγικές που θα αναπτύξουμε για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές πραγματικότητες. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά και οι στρατηγικές κατάρτισης εδώ καλούνται να καλύψουν τα κενά αυτά. κουλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' θα ήθελα να πω πως είναι καλή η γνωμοδότηση. Ναι, σωστό να αποδίδουμε την κατάλληλη σημασία στην εκπαιδευτική κατάρτιση. Είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά έχω την αίσθηση πως ε, πρέπει να έχουμε κατά νου την ε, γενικότερη εικόνα και το ευρύτερο πλαίσιο ίσως κάπως οι δομές να είναι πολύ άκαμπτες. Θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Έχω συνεργαστεί και με τον τομέα τον δημιουργικό με δύο επιχειρήσεις. Η ε, ε, μία είχε 30 εργαζόμενους και τώρα έχει φτάσει στους 60. Ε, και ήθελα να δραστηριοποιηθεί στην Ισπανία. Αλλά το πρόβλημα ποιο ήταν. Τους προσέφεραν οι Αμερικανοί 5 εκατομμύρια για να εγκατασταθούν εκεί πέρα, 100 εκατομμύρια οι Κινέζοι για να πάνε στην Κίνα, οπότε δεν είναι τίφτο το ζήτημα εναλλακτική. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αναζητήσουμε κάποιους ε, συμβούλους για να εργαστούν για αυτή την ε, εταιρεία για να αντλήσουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα ήταν 3-4 εκατομμύρια. Και ξέρετε πως αυτό οδηγεί στο ότι οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται φεύγουν. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε οι επιχειρήσεις ε, που αναπτύσσονται να έχουν εδώ πέρα τις απαραίτητες προϋποθέσεις ε, και τις τράπεζες που χρειάζονται και τη χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα προβλήματα στον τομέα των δημιουργικών που απασχολεί νέους. Και φοβάμαι πως έτσι δεν θα μπορέσουν ε, να προσφέρουν, δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν θέσεις εργασίας. Το μόνο που θα απομείνει θα είναι στήριξη, επιδόματα κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να ε, παραμείνει εδώ πέρα η τεχνογνωσία η οποία αναπτύσσεται. Γι' αυτό ε, ανασυχώ για, την, ε, το γενικότερο πλαίσιο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Δεν θα επιτύχει αυτό εάν δεν μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις που έχουν ανάπτυξη και θα ήθελα να μείνουν εδώ. Εν ολίγης, αυτά τα οποία πρότεινε είναι σημαντικά πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα, ε, τη γενικότερη εικόνα. Όλοι μαζί, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για να ε, δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα στον τομέα αυτόν. Ευχαριστώ, Ταβάρες. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα περισσότερα από αυτά τα σημεία αναφέρθηκαν ήδη. Τα δύο αυτά θέματα συνδέονται. Εγώ θα αναφερθώ στη χρηματοδότηση και θέλω να επισημάνω πως παρά το ότι οι δηλώσεις καλής πίστης και συνεργασίας από τα άλλα κράτη-μέλη είναι ευπρόσδεκτες, σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη και αυτά τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Από όταν ξεκίνησε η κρίση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει στις χώρες της ε, κρίσης ε, ατυχής, ε, τις λεγόμενες pigs, αλλά σε επίπεδο χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα πριν την κρίση και χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα έπρεπε να επενδύει περισσότερο εκεί πέρα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το εξηγεί λέγοντας πως πρέπει να διατηρήσει το 3α τη δική της αξιολόγηση και άρα δεν μπορεί να επενδύσει στις χώρες της κρίσης όπως ε, στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της σύσταση μιας υπηρεσίας της Ένωσης για έργα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. που θα είχε υψηλότερη αξιολόγηση από την Ελλάδα και την Πορτογαλία και θα μπορούσε να επενδύσει σε έργα προσθέμενης αξίας για το μέλλον στις χώρες της ε, κρίσης και νομίζω πως θα λειτουργούσε ως αντίβαρο στην ε, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση Πορτογαλίας, Ιταλίας και λοιπόν χωρών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο να προσθέσω. Νομίζω πως η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ θετική και μπορούμε σε γενικές γραμμές να τη στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Εκτιμώ πολύ την έκθεση που ετοίμασε ο εισηγητής μας, διότι πιστεύω ότι όπως αναφερόταν και πριν, η εφετηρία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι ένα καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης. Έχουμε μια χώρα που υπάρχει ανεργία των νέων που σπάει ρεκόρ και το σύστημα της παιδείας είναι σύστημα που δεν είναι ιδιαίτερα καλό το επίπεδο ποιότητας του Πανεπιστημίου του Ιταλικού όσον αφορά την προετοιμασία για την εργασία των νέων μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλή βαθμολογία. Άρα χρειάζεται σίγουρα μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ προετοιμασίας πανεπιστημιακής κατάρτισης εν γέννη και του κόσμου της εργασίας. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλούς τέλειους ε, επαγγελματίες στον τομέα των επικοινωνιών παραγματος χάρη, για να πάρουμε ένα παράδειγμα των επιστημών, ε, το παράδειγμα του αλληλικού, χωρίς να υπάρχουν ανάλογες θέσεις εργαστούν αυτοί οι νέοι που έχουν αυτά τα προσόντα. Και χρειάζεται και το διπλό σύστημα, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα μαζί με τις σπουδέ να προωθείται μαζί με τη θεωρία και η πρακτική. Ε, και σε αυτό βλέπω τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και της προετοιμασίας ενός πτυχιούχου στην ε, νομική Ιταλού, ίσως και σε άλλες χώρες, και εκείνον που θέλει να κάνει το δικηγόρο και δεν βλέπει πριν πάρει το πτυχίο κάνει το δικαστήριο. Ίσως σε σχέση με άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες και με τη ΣΥΠΑ υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι θεμελιώδες σημείο. Πρέπει να υπογραμμιστεί και να συμπληρωθεί το θέμα των κινήτρων για τους νέους. Δηλαδή σε πολλές χώρες υπάρχουν συστήματα φορολογικά, υπερβολική φορολόγηση, πολύ βαρύς φόρος, που πολύ συχνά εμποδίζει τους πιο νέους να ανοίξει επιχείρηση, ε, να μπει στην αγορά εργασίας, να μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή την καριέρα του. Διότι υπάρχει φορολόγηση που δεν βραβεύει το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων. Άρα σε περίοδο λιτότητας και κρίσης όπου οι χώρες ε, επιβάλλουν πολύ σοβαρές φορολογικές θυσίες εκείνοι που δέχονται μεγαλύτερο ε, βάρος οι νέοι που δεν μπορούν να επενδύσουν αλλά έχουν μεγάλη φαντασία, ε, έχουν την επιθυμία να εργαστούν αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στον κόσμο εργασίας λόγω των μεγάλων φόρων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσε να συμπληρωθεί σε αυτά που παρουσιάζει η έκθεση. Αυτές μπορούν να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της δουλειάς που θα κάνουμε και εδώ, αυτές που αναφέρθηκαν και συζητούνται. Ευχαριστώ. Κύριος Καβαντά. Ευχαριστώ. Έχω τέσσερις παρατηρήσεις γρήγορες και ένα σχόλιο που απευθύνεται προς τον κύριο Ντελβάη. Εξεπλάγει. Μάλλον ε, με συγκλώνησε η έξοχη ποιότητα της, της λογικής που ακολουθήσατε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ρεαλιστική η προσέγγισή σας και πίσω από όλα αυτά βλέπουμε τη μακρά εμπειρία στο δημόσιο βίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία. Λοιπόν, η ενεργεία των νέων, πρώτη παρατήρηση. Ε, καταρχάς, όπως είπε, αναφέρθηκε πρόσφατα ο συνάδελφος ο κ. Σκορία, που τα ανέφερε, αφορά το θέμα της παιδείας. Εκεί πρέπει να κινηθούμε, στον τομέα της παιδείας κατεπηγόντως, διότι σε κάποιες χώρε. Έχουμε συστήματα απειρχαιωμένα που δεν είναι προσαρμοσμένα στις συζητήσεις της οικονομίας και αυτό είναι κάτι που αυξάνει την ανεργία των νέων. Δεύτερη παρατήρηση, δεύτερο σχόλιο, η δουλειά των νέων δεν απομονώνεται από το, από το υπόλοιπο οικονομικό πλαίσιο. Η εργασία των νέων είναι πιο ικανοποιητικά, ικανοποιητικά αν υπάρχει ε, ανάπτυξη, δηλαδή υπάρχει ζήτηση, χρειάζεται μια μεταρρύθμιση του πλαισίου της εργασίας, αλλά θα πρέπει να τονώσουμε παντιοτρόπος μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στα προϊόντα που σκευάζουμε και παραδίδουμε, διότι μιλάμε για μια παγκόσμια αγορά στην οποία κινούμαστε. Τρίτη παρατήρηση. Θα πρέπει, και όλοι αρχίζουν να το αισθάνονται αυτό, θα πρέπει να έχουμε σοβαρές δημοσιονομικές ε, πολιτικές, αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε τις ζημιές που προξανεί η λιτότητα. Πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Χρειάζεται σοβαρή ευρωπαϊκή κυβέρνηση γι' αυτό, με μέσα συγκεντρωμένα και όχι εξουδετερωμένα. Και το τέταρτο σχόλιο μου εξ αυτού. Από το 2008 βλέπουμε έλλειψη πολιτικής διακυβέρνησης της οικονομίας, της νομισματικής οικονομίας, της φορολογίας και του κοινωνικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και υπάρχει αδράνεια των συστημάτων. Όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν. Διότι η κρίση είναι ανεφροηγουμένου. Ποτέ δεν είδαμε από δεκαετία του 30 στην Ευρώπη πάνω από το μισό των νέων σε κάποιες χώρες να μην έχει πρόσβαση στη δουλειά. 30 ε, με 32 χρόνια. Εμείς βασιζόμαστε, μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε. Θα πρέπει να είναι πιο ισχυρή η φωνή μας, ε, να ξυπνήσουμε τους θεσμούς. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι προσπάθειες σε πολιτική ενότητα, μια διακυβέρνηση οικονομική και θα πρέπει να υπάρξουν συστήματα που λειτουργούν και να λειτουργούν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά που έλεγε ο κ. Σταβάρε, ακούσαμε ότι υπάρχουν δυσκολίε στι Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πιστεύουμε ότι ονειρευόμαστε. Δηλαδή, η τράπεζα φοβάται να δανειστεί για να μην χάσει τη βαθμολογία τη και να μην είναι αξιόπιστη στο, ε, στην αγορά την πιστοληπτική. Θα πρέπει οι πολιτικοί να κάνουν τη δουλειά τους. Θα πρέπει να ηγηθούν, να κατευθύνουν, να δικήσουν οι πολιτικοί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παναγιώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Μενέντε Δεβάγε για την προσπάθεια που έκανε και για τις συστάσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης για να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες mm. μεταρρύθμισης στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία συγκεκριμένα σημεία που έχουν την δυνατότητα να συναποτελέσουν, θα έλεγα, τμήμα του εγγράφου μας. Πρώτον, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Έτσι το διδακτικό σώμα θα έλεγα θα πρέπει να αναπτύξει καινοτόμες δράσεις διδασκαλίας και εκμάθησης. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που με τη σειρά τους θα τους επιτρέψουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να ανοίξουν νέες προοπτικές απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης ε, να συνδέσουμε την εκπαίδευση, της επιστήμες και την επιχειρηματικότητα στις χώρες μας. Έτσι, ε, αν δεν προχωρήσουμε, κάθε έξι μήνες θα προσθέτουμε 200.000 νέους ανέργους και θα πρέπει να προωθήσουμε την εκμάθηση αρμοδιοτήτων και γνώσεων και ικανοτήτων σε τομείς όπως η έρευνα και η πληροφορική εκεί που έχουμε ελλείψεις. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη μέσω των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων θα πρέπει να προωθήσουν τον τομέα αυτό της πληροφορικής και, και των μαθηματικών. Θα πρέπει επίσης η Ευρώπη να πάρει μέτρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους. Έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις που υπάρχουν και να απομακρύνουμε τον φόβο της αποτυχίας στους νέους, οι οποίοι πιστεύουν ότι αν δεν πετύχουν δεν θα μπορέσουν να εργαστούν. Κλείνοντας να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις διαρκής. Ο νέος δεν θα πρέπει απλά να βλέπει και να εκμεταλλεύεται αυτά που του προτείνουμε, αλλά να πάρει μέρος στις διαδικασίες, ε, θα έλεγα, διαμόρφωσης των μέτρων που αφορούν την εκπαίδευσή του. Σαντιάγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ντελβάγε έχει δώσει μια συγκεκριμένη θα έλεγα εικόνα του πώς έχουν τα πράγματα. Στον τομέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εγώ είμαι πρωταγωνιστής για αλλαγές στον τομέα της παιδείας στην Ισπανία. Έχω την αίσθηση και το έχω επαναλάβει αυτό ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε την πολύ μεγάλη αξία και σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Αυτό έχει πολύ μεγάλη επαναλαμβάνω σημασία. Να επανέλθω σε κάτι που έθεσαν άλλοι συνάδελφοι και να κάνω μια πρόταση προς τον Εμίλιο. Θα πρέπει να στηρίξουμε επίσης με συγκεκριμένο τρόπο και τους νέους που είναι νέοι επιχειρηματίες. Πολλές φορές οι νέοι στην Ισπανία στοχεύουν να γίνουν υπάλληλοι, να εργαστούν σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, σε τράπεζες και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες, το είπε και η συνάδελφος Παναγιώτοδα και θα πρέπει να, να καταλάβουμε ότι η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας είναι αυτοί που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε γενικά την επιχείρηση. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά γραφειοκρατικά βάρη για την δημιουργία μιας επιχείρησης, κάτι το οποίο στη δική μου χώρα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και βαρύ. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Είναι η κατάλληλη εργατική νομοθεσία, το έθεσε και η Μίλανα. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της πτώσης της απασχόλησης των νέων προέρχεται από την εργατική νομοθεσία. Στη δικτατορία του Φράνκο οι εργαζόμενοι δεν είχαν δικαιώματα θεμελιώδη. Δεν είχαν το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε, δεν είχαν το δικαίωμα του απεργήν. Αυτά τα απέκτησαν αργότερα, αλλά ήδη από την εποχή του Φράνκο ο ε, εργαζόμενος ήταν υπερπροστατευόμενος. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον απολύσουν. Ήταν καταστροφικό για τις ε, επιχειρήσεις. Περάσαμε τώρα από αυτή την κατάσταση σε μια νέα σειρά συμβάσεων για τους νέους έξι μηνών και όταν ήλθαν, ήλθαν οι δύσκολοι καιροί, ήρθε η οικονομική κρίση, τότε προχωρήσαμε ε, σε καταστάσεις οι οποίες ε, είναι ιδιαίτερα απογοητευτικές για τους νέους. Η έλλειψη θέσεων απασχόλησης στην Ισπανία ε, δεν είναι τόσο δραματική. Αυτό που είναι δραματική είναι η κατάσταση των νέων που έχουν μερικές φορές συμβάσεις εργασίας ιδιαίτερα περιορισμένες χρονικά και αφού εργαστούν λίγο βρίσκονται μετά σε μια παράδεκτη κατάσταση και είναι πάρα πολλοί που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση και μόνο μια βελτίωση της οικονομίας θα τους βοηθήσει. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχουν συστήματα όπως στην Δανία ο Μόρτεν μπορεί να μας βοηθήσει της ευελιξίας της ε, των εργασιακών ρυθμίσεων που θα μπορέσει, επαναλαμβάνω, να ε, βοηθήσει ιδιαίτερα. Ο κύριος Τόμας βάνε από την Κομισιόν, σωστά το είπα, δεν είναι εκεί. Κυρία μου, δεν ξέρω το όνομά σας. Τέσσερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φιωρέλα Περότο από την Γενική Διεθνής Εκπαίδευση και Πολιτισμού. Ναι βεβαίως συμφωνούμε με το περιεχόμενο του σχεδίου γνωμοδότησης και δεκτές και οι συστάσεις της Επιτροπής που εντοπίζουν τους τομείς όπου χρειάζεται δράση. Και συγκεκριμένα συμφωνούμε με την πεποίθηση πως η εκπαίδευση και η κατάρτιση παίζουν ένα ρόλο κλειδί στη μείωση και πρόληψη της ανεργίας των νέων και είναι πράγματι καλύτερη ασφάλεια θα έλεγε κανείς κατά της ανεργίας των νέων. Καλωσορίσουμε επίσης την έμφαση που δίνεται στην ανάγκη να μειωθεί η εγκατάλειψη του σχολείου και να προληφθεί το φαινόμενο ως ε, ένας βασικός τρόπος να μειωθεί η ανεργία των νέων, ειδικά σε τομείς ε, και ομάδες νέων ε, όπου έχουμε πολλούς νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο επίσης. Σημαντικό είναι ότι ο συγητής ε, τονίζει το ζήτημα της κινητικότητας στη μάθηση για να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των νέων, αλλά και άλλα ζητήματα όπως ε, εγκάρσιες δεξιότητες και δεξιότητες κλειδιά, όπως παραδείγματος χάρη γλώσσες, αλλά όχι μόνο αυτές και επίσης η σημασία που έχει χρήση του νέου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για να αυξηθεί η μαθησιακή κινητικότητα. Επίσης συμφωνούμε πλήρως με την ανησυχία σας για τις απειλές του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση και κατάρτιση και τις περικοπές. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν ζήτησε από τα κράτη-μέλη να κάνουν μια διαφορετική εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, κάτι οποίο σημαίνει πώς ε, θα ε, δώσουν μια διαφορετική προτεραιότητα στην εκπαίδευση και στην ε, κατάρτιση. Επίσης, στην ανακοίνωση τη σχετική, εμείς προτείναμε να ξεκινήσουν συζητήσεις στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με τα κράτη-μέλη για την χρηματοδότηση των συστημάτων αυτών και, στη, και για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Ειδικά σε καιρούς ε, δύσκολους για να διατηρηθεί και να αυξηθεί η ποιότητα. Επίσης συμφωνούμε με την ανησυχία σας και την έκκληση που γίνεται να ενισχυθεί η μάθηση στον χώρο εργασίας για να είναι πιο επίκαιρες οι δεξιότητες, πιο κοντά στις ανάγκες αγοράς εργασίας, να μειωθεί η... το ότι δεν είναι οι δεξιότητες αυτές οι οποίες ζητάει η αγορά και επίσης βεβαίως να δούμε και την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, όχι μόνο της επαγγελματική ε, κατάρτισης, για να υπάρχει και αριστεία και μεγαλύτερη απασχολησιμότητα. Και η ποιότητα πράγματι είναι ένα σημαντικό κομμάτι του εξυγχρονισμού της ανώτατης εκπαίδευσης ε, που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά της Κομισιόν με τα κράτη-μέλη. Επίσης, μιλάτε για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών ε, μέσων για τη διαφάνεια και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων γιατί έτσι θα ενισχυθεί η κινητικότητα στον κλάδο αυτό για να μπορέσουν τα προσόντα να είναι αυτά τα οποία ζητάει η, εργασία, η αγορά εργασίας και να αυξηθεί η απασχολησιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι βεβαίως ε, δίνεται αξία και στο αποτέλεσμα άτυπης ε, ή ανεπίσημης εκπαίδευσης πράγματα τα οποία τονίσαμε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης. Καλώς ορίζουμε επίσης την έκκληση που απευθύνουν στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του... της εγγύησης για τους νέους μέσω υπαρκούς χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την εστίαση ιδιαίτερα στις περιφέρειες και τις ομάδες που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Και αυτό νομίζω προέκυψε συζήτηση. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω πως αύριο 29 Μαΐου η Κομισιόν θα υιοθετήσει τις ε, συστάσεις αναχώρα και οπωσδήποτε πολλές από αυτές τις συστάσεις θα αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που είχε αναφέρει η Κομισιόν. Θα Σταματήσω εγώ εδώ, είναι και συνάδελφός μου, δεν ξέρω αν θα θέλετε να προσθέσετε κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Νομίζω πως δεν υπάρχουν πάρα πολλά να προσθέσουμε. Ποιος είναι. Όχι. Εντάξει, ωραία. Δεν ναι, θέλετε το λόγο. Χαίρομαι. Να δώσω λόγο στον κύριο Ντελβάλε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς. Ίσως να υπήρξε και μία κάποια μικρή παρανόηση και θα ήθελα να το διευκρινίσω. Εγώ τέλειωσα την παρέμβασή μου λέγοντας ότι συμφωνώ μαζί σας, ότι βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο εδώ. Επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εγώ αναφέρθηκα επίσης και στα εμπόδια τα κοινοβουλευτικά τα οποία μπορούμε να, συνεχί, να συναντήσουμε στα πλαίσια της έγκρισης από την Ομοσπονδιακή Βουλή. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την πρωτοβουλία της Κακελαρίας. Απλά επαναλαμβάνω ότι είναι μια προφανής δημοκρατική θα έλεγα προϋπόθεση, άβολη στη συγκεκριμένη περίπτωση, να εξεταστεί η πρόταση αυτή και από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή και αναφέρθηκα ακριβώς στην πιθανή λυπηρή θα έλεγα καθυστέρηση ε, γιατί ε, στην ουσία η πρόταση θα εφαρμοστεί μόνο μετά τις εκλογές. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στην ομοφωνία η οποία υπάρχει, στη συνένεση να το πω καλύτερα, όλων των ιδεολογικών απόψεων που αντιπροσωπεύονται εδώ. Θα ήταν πραγματικά παράλογο να υιοθετήσουμε μέτρα να μην υιοθετήσουμε μέτρα τα οποία ε, θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ανάκαμψη της απασχόλησης στους νέους. Τα σχόλια λοιπόν τα οποία έγιναν από ορισμένου ε, βουλευτές, συναδέλφους, άνδρες και γυναίκες, κάποιοι έχουν ε, φύγει αυτή τη στιγμή. Θα συμφωνήσω κυρίως με αυτά τα οποία είπε η κυρία Σάντσες Σμιτ ο κύριος Στακούλα είναι εδώ και συμμερίζομαι και με αυτά τα οποία είπε. Απαιτείται να υπάρξει μια συνένεση για τον κύριο Ταβάρες. Πράγματι το θέμα της χρηματοδότησης είναι το κυρίαρχο. Και το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια ότι ε, δεν θα πρέπει να αποκρύψουμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. και θα μπορέσετε αν θέλετε να το θέσετε το θέμα αυτό και με τροπολογίες και με συμβιβαστικών τροπολογιών να υπάρξει αυτή η πιθανή υποδιέρεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι μια ιδέα η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά. Για τον κύριο Σκουρία, ε, πράγματι η βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων της παιδείας της χώρες είναι απαραίτητο. Το σύστημα αυτό το διπλό το οποίο εφαρμόζεται είναι εν γνώση όλων μας και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν στους νέους και μέσω των φορολογικών μέτρων, το οποίο έθεσε ξεκάθαρα και ο κύριος Φίσας. Σήμερα πάρα σε πάρα πολλές χώρες οι φορολογικές ρυθμίσεις δεν ευνοούν τους νέους επιχειρηματίες. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε έτσι ώστε να γίνει αυτό στην κυρία Τομά. Ε, εκφράζω τη συμφωνία μου με αυτά τα οποία είπε. Δεν μπορούμε βέβαια μόνο να αντιμετωπίσουμε τους νέους σαν ένα μεμονωμένο πεδίο πειραματισμού. Ε, πρέπει να δούμε τα προβλήματά τους σε σχέση και με τα προβλήματα του συνόλου των εργαζομένων. Να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Καβαντά για την έλλειψη της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία καλούμεθα να συζητήσουμε σήμερα. Μετά από 60 χρόνια να βρισκόμαστε στην κατάσταση να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει έλλειψη οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι λυπηρό. Θα συμφωνήσω επίσης και με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ταβάρες λίγο πιο πριν ότι πραγματικά είναι, δεν θα πρέπει να προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες της και να μην χρηματοδοτεί μόνο και μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να μην διακινδυνεύσει τη σωστή της βαθμολογία, την καλή της βαθμολογία. Και για την κυρία Παναγιώτοβα να πω ότι αυτά που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και να επίσης μια λεπτομέρεια θα έλεγα εγώ έχω πάρα πολλούς καθηγητές και δασκάλους στην οικογένεια. Προφανώς, προφανώς και θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες εξελίξεις και να υιοθετήσουν τις νέες μεθόδους. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν να αναπτύξουμε επίσης και το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων να διευκολύνουμε την απασχολησιμότητα των νέων αυτών και μέσω φορολογικών ρυθμίσεων που να ευνοούν τους νέους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα θα μειωθούν. Να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο φίλος Σαντιάγο Φίσας ότι η μεταρρύθμιση των εργασιακών ρυθμίσεων ε, είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει. Ε, αυτά τα οποία συνέβαιναν την εποχή του Φράγκο είναι χρήσιμο να σημειωθεί τι αποτελέσματα είχαν, θα έλεγα, δημιουργήσει, που μας είχαν οδηγήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεβάγιο. Ένα θέμα δεν αναφέρθηκε. Δεν λέτε τίποτα για το ζήτημα της αποταμίευσης. Να δείτε πώς οι νέοι οι Γερμανοί θα μπορούσαν να δουλέψουν Και δεν μπορούν να το κάνουν γιατί, γιατί δεν ξέρουν τη γλώσσα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές λοιπόν οι γλώσσες. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη χώρα όπως η Γερμανία που έχει θέσεις εργασίας και έχει κακή δημογραφική κατάσταση, νομίζω καλό θα ήταν ε, να σκεφτεί κανείς θα μάθω γερμανικά γιατί εκεί πέρα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Όχι για να φύγει από την ε, Ισπανία αλλά για να μπει κάπως στην αγορά εργασίας. Αυτά λοιπόν για το θέμα των ε, γλώσσων. Λοιπόν, 5η, 12 η ώρα, οι τροπολογίες ε, λύεται τη συνεδρίαση τώρα, γιατί θα ακολουθήσει η συνεδρία των συντονιστών. Ξεκινάμε 3,5 ώρα με τις ψηφοφορίες. Εντάξει, 3 και μισή. Λοιπόν, Βγείτε παρακαλώ από την αίθουσα για να συνεδριάσουν οι συντονιστές. Yeah,